Uh, good morning, colleagues and uh, other friends. I'm tempted to start the meeting because we have a tough agenda, and um, uh, I could uh, give my uh, chairman. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να ξεκινήσω τώρα τη συνεδρίαση. Γιατί έχουμε αρκετά φορτωμένη μερή σε διάταξη. Στο μεταξύ θα έρθουν και οι συνάδελφοι σιγά-σιγά. Θα πρότεινα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας. Στο σημείο 1, συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Μία αλλαγή προτείνω μόνο. Η συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Αυτό ζήτησε ο Πρόεδρος. Ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση. Έλεγα να αρχίσουμε πρώτα το το αργότερο 10 παρατέταρτο την ακρόαση για την Ανατολική Ασία, γιατί έχουμε και άλλη σημαντική ακρόαση με την Κίνα, που θα πρέπει να αρχίσει το αργότερο στι 11, οπότε δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 26 και 27 Απριλίου του 2010. Μπορούμε να τα εγκριμε ωραία. 10 Μαΐου του 2010 και δεύτερη και τρίτη Ιουνίου του 2010. Εγκρίνονται τα πρακτικά των τριών συνεδριάσεων. Σημείο 3. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Θα ήθελα στις θερινές σας διακοπές να σκεφτείτε τον επόμενο βραβευθέντα το, για το βραβείο Ζαχάροφ, γιατί οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν πριν τις 6 το απόγευμα στις 22 Σεπτεμβρίου. Και όπως ξέρετε, οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε από πολιτικές ομάδες είτε από 40 ε, το λιγότερο μεμονωμένων ευρωβουλευτών. Και θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε το επόμενο βήμα μετά την υποβολή των υποψηφιωτήτων θα είναι στις 5 Οκτωβρίου σε κοινή επιτροπή των, επιτροπών σε κοινή συνεδρίαση των Υποεπιτροπών ανάπτυξη Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε αυτή την κοινή συνεδρίαση θα υποβληθούν οι υποψηφιότητε για το βραβείο Ζαχάροφ και η ψηφοφορία για τους τρει ε, επικρατέστερου θα γίνει από τη κοινή συνεδρίαση πάλι των τριών επιτροπών στι 12 όμω Οκτωβρίου. Εκεί θα διαλέξουμε έναν από του τρει τελευταίους ε, επικρατέστερο υποψήφιο. Αυτά να τα έχετε υπόψη για να σκεφτείτε τον επόμενο υποψήφιο. Σήμερα έχουμε την 15η Ιουλίου. Πέρυσι την ίδια μέρα είχαμε τα εγγένεια της νέας ε, κοινοβουλευτικής θητείας, αλλά μάθαμε και τα θλιβερά νέα της ε, δολοφονίας της Νατάλιας Στεμίραβα. Μάλιστα μας συγκλώνησε αυτό το γεγονός και ίσως επηρέασε την περσινή απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Και πραγματικά είναι πολύ ατυχές που μέχρι στιγμής δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία αυτή. Μάλιστα το Memorial, η Ένωση Memorial, εξακολουθεί να υφίσταται παρενοχλήσεις από τις ρωσικές αρχές. Μάλιστα ο πρόεδρος Μπούζεκ ε, εξέδωσε και μια ανακοίνωση ε, επ' ευκαιρία της πρώτης επαιτίου από τη δολοφονία της Νατάσα Στεμίροβα. Επίσης θα διαπιστώσετε ότι ε, στις 12 Ιουλίου καταδικάστηκαν ε, δύο ε, αντιρρησίες, ένας από το Μουσείο του Βραβείου Ζαχάροφ και ένας καλλιτέχνης σε πρόστιμα 150.000 και 200.000 ρουβλίων αντίστοιχα για μια ε, οργάνωση απαγορευμένης έκθεσης. Μάλιστα, ο εισαγγελέα θεώρησε ότι δύο κατηγορούμενοι είχαν ε, χρησιμοποιήσει ως τα εκθέματα θρησκευτικά σύμβολα με τρόπο να υποδαβλίζουν ε, τη μυσαλλοδοξία, και υπονομεύοντας ε, την εικόνα των Ορθόδοξων Χριστιανών. Παρακολουθήσαμε αυτή τη δίκη στη Μόσχα με πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις και κατά πάσα πιθανότητα οι δύο κατηγορούμενοι, Γερόβιεφ και Σαμόντοροφ, θα ασκήσουν προσφυγή, θα υποβάλουν έφεση. Και μάλιστα ο πρόεδρος της, κοινής, ε, της Μικτής Κοινοβουλευτικής Αποτροπής, ο κ. Φλέκεστάιν, ε, Ξέδωσε και ανακοίνωση για τη δικαστική αυτή απόφαση, εκφράζοντας ε, την επιθυμία του να συναντήσει τους δύο καταδικαστέντες την επόμενη φορά που θα μεταβεί στη Μόσχα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι μετά την απόφαση για το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής μια τριμελής αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Μπίεσλαν της Ρωσίας, στην Νότια Οσετία, για, τον για την εκδήλωση αυτής της τραγεδίας, τότε που πάνω από 100 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια αντιτρομοκρατική δράση. Η τριμελής αυτή αντιπροσωπεία παρτίζεται από την υποφαινόμενη, την αντιπρόεδρο Αντρικένε και τον κύριο Μπέρμαν. Εμείς οι τρεις λοιπόν θα πάμε στο Μπίεσλαν για την εκδήλωση αυτή, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. και με οικογένειες των θυμάτων την 1η Σεπτεμβρίου. Η... Τα επίσημα εγγένεια του δικτύου Ζαχάροφ, τον πρόεδρο Πέτερινγκ το 2008, είχε μια συνέχεια. Επιτέλους το Προεδρείο υιοθέτησε ένα σημείωμα για τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας αυτού του δικτύου Ζαχάροφ. Απόφαση προβλέπει ότι το δίκτυο αυτό θα υποβάλει κοινέ εκκλήσει, θα οργανώνει αντιπροσωπείε, θα συνεδριάσει μεταξύ των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπείων και των βραβευθέντων βραβείο Ζαχάροφ στι χώρε προέλευσή του. Επίση, θα προσκαλεί βραβευθέντε σε εκδηλώσει, θα οργανώνει επίσης διαλέξεις σε σημαντικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής το δίκτυο αυτό θα συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο τελευταίος βραβευτής με το βραβείο Ζαχάροφ. Επόμενο θέμα, η Σρι Λάγκα. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτά που συμβαίνουν στη Σρι Λάγκα αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει το γεγονός, το, το καθεστώς ε, γενικευμένο προτιμήσω ΣΥΝ προς το καθεστώς της Σρι Λάγκα, γιατί η κυβέρνηση δεν ε, έδειξε προθυμία να τηρήσει τις 20 ε, ερήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου οι εμπορικέ παραχωρήσει να παραταθούν για ένα εξάμεινο ακόμη. Δεν τηρήθηκαν αυτέ οι 20 υποχρεώσει από το Σρι και ανέστηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση του GSP+. Για τη Συρία. Με μεγάλη απογοήτευση ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα το σημαντικό υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριο Αλμάλη, δικηγόρο στο επάγγελμα, καταδικάστηκε σε Συριακό στρατοδικείο στις 4 Ιουλίου σε τριετή φυλάκιση με, κατηγορία την ε, διάδοση ψευδών ειδήσεων ε, για τη Συρία προκειμένου να υπονομεύσει το ηθικό του έθνους. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ε, αιτιολογικά διατακτικά αποφάσεων είναι τόσο αόριστα και αφηρημένα. Πραγματικά μα δημιουργούν τεράστια θλίψη γιατί ο κύριος αυτός είναι 79 ετών, ήδη ασθενή και θα προσπαθήσουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε, αυτό σε αυτή την κατάσταση προκειμένου να ανασταλεί η πίνη του. Άλλωστε θα εφεσιβληθεί και η απόφαση. Συνήθως ζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις ε, ακόμη και αν είναι στη φυλακή, να έχει πρόσβαση σε τροφαρμακευτική περίθαλψη και να τύχει σωστή μεταχείριση. Ελπίζουμε ότι οι Συριακέ Αρχέ θα βρουν ένα ευφύ τρόπο για να αναστείλουν την φυλάκιση του, την έκθεση τη ποινή του. Πραγματικά δεν ε, ε, είναι μια τιμή για τη Συριανή δικαιοσύνη. Είχαμε στι 10 Ιουλίου μια ακρόαση για την πολιτική γειτνία. Μετά την παρουσίαση του Μωάτε Σελφετζήρη, η Αιγυπτιακή εφημερίδα Λαχράμ στις 22 Μαΐου εξέδωσε ένα άρθρο ε, με, κα, με κατηγορίες κατά του δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στις Βρυξέλλες για τις επικρίσεις που άσκησαν στην Αίγυπτο για την αντιμετώπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κρίμα που απαγγέλθηκαν τέτοιες κατηγορίες από μια εφημερίδα που πρόσκειται ουσιαστικά στην κυβέρνηση τη Αιγύπτου. Την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκαν τρία κατεπήγοντα ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στην Κυργυζία, Κυργιστάν. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τα πρόσφατα γεγονότα και με παρουσίαση και διεθνών προσώπων αν γίνεται και παρατηρητών. Επίσης ζητήσαμε η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνοδευτεί από προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασης και αποτροπή της επανάληψης της βίας. Η απειλή αυτή εξακολουθεί να υπάρχει και μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια και την ειρήνη και στις γειτονικά Ταζικιστάν και Ουσμπεκιστάν. Το τρίτο ψήφισμα αφορούσε τη Βόρεια Κορέα. Στο ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για την απογοητευτική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και το ψήφισμα αυτό συνεχίστηκε από μια πολύ σημαντική ακρόαση που διοργανώσαμε εμείς στην Επιτροπή μας πριν από μερικούς μήνες. Το ψήφισμα αυτό καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να Υποβάλλουν ένα ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητώντας από τη Βόρεια Κορέα α, να, τα εγκλήματα που έγιναν εκεί να δικαστούν σε διεθνές δικαστήριο συμπεριλαμβανομένων των εξοδικαστικών α, εκτελέσεων των στρατοπέδων φυλακισμένων και το καθεξής. Επίσης, ζητούμε την συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής στα Ηνωμένα Έθνη για να εξετάσει την κατάσταση παραβίας δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ειδικό απεσταλμένο στη Βόρεια Κορέα. Αυτό ήταν στο δεύτερο ψήφισμα. Το τρίτο ψήφισμα αφορούσε την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Ήταν κατεπήγον ψήφισμα για την περίπτωση του Φαράι Μαγκούμπου, του ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μίλησε ανοιχτά για καταστρατηγής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα δαματορυχεία της Ζιμπάμπουε. Τελικά του δόθηκε, βγήκε με εγγύηση τον Ιούλιο μετά από ένα μήνα φυλάκισης, αλλά εξακολουθεί να κατηγορείται για δημοσίευση και ανακοίνωση ψευδών πληροφοριών που βαίνουν, βάλουν κατά του κράτους. Βλέπετε παρόμοια η απαγγελία κατηγορίας με αυτή που έγινε στη Συρία. Δεν είναι οι μόνες χώρες βέβαια που έχουν στο ποινικό τους δίκαιο τέτοιες αόριστες, τόσο αόριστα τυποποιημένα εγκλήματα. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον ακτιβίστη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ζιμπάμπουε. Μια άλλη σημαντική είδηση είναι ότι η κουβανική κυβέρνηση πρόσφατα απελευθέρωσε μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων. Οι πολιτικοί αυτοί κρατουμένοι και οι οικογένειές τους ε, εξορίστηκαν στην Ισπανία. Μεταξύ τους βρίσκονται και, τα, και οι συγγενείς των γυναικών ε, με τα του που έχει βραβευθεί με το βραβείο Ζαχάροφ πρόσφατα αυτή η ένωση και μάλιστα ο πρόεδρος Μπούζεκ είπε ότι οι αρχές αρχίζουν ε, να λαμβάνουν πιο σοβαρά υπόψη αυτή την απεγνωσμένη έκκληση που έγινε για την ελευθερία έκφρασης. Η υποεπιτροπή μας θα οργανώσει μια ανταλλαγή απόψεως στις 8 Νοεμβρίου με θέμα την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και θα έχουμε συνεχή επαφή μεταξύ του γραφείου του Πρόεδρου Μπούζεκ και της Ένωσης Γυναίκες στα Λευκά για να δούμε αν μπορούμε να προσκαλέσουμε εκπροσώπους της στην Ολομέλεια προκειμένου να μπορέσει αυτή η οργάνωση να λάβει το βραβείο Ζαχάροφ που της έχει απονεμηθεί στο Στρασβούργο σε επίσημη τελετή. Αυτές είναι ανακοινώσεις προς το παρόν, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί δεν μας περισσεύει ο χρόνος σήμερα. Α, μόλις ε, έλαβα και μία επιστολή από τον ε, Γενικό Εισαγγελέα Λουίς Μορένο Κάμπο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα θυμάστε ότι τον είχαμε καλέσει στην Επιτροπή μας πριν από λίγους μήνες. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τις επαφές που είχαμε και επίσης ε, φυστά την προσοχή μας σε μία απόφαση προδικαστική της 12ης Ιουλίου για τον Ομάρ Αλμπασίρ, τον πρόεδρο του Σουδάν. Και λέει ότι το προδικαστικό συμβούλιο εξέδωσε και δεύτερο ένταλμα σύλληψης κατά του πρόεδρου Αλμπασίρ, στην περίπτωση αυτή για τρεις κατηγορίες γενοκτονίας. Και μάλιστα ο επικεφαλής αγγελέας, ο κ. Μορένο Κάμπο, ε, εκφράζει την ελπίδα ότι μια και το έγκλημα της γενοκτονίας είναι το πιο σοβαρό έγκλημα με βάση το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, ελπίζει ότι θα τον βοηθήσουμε στην προσπάθεια να προσαχθεί ο πρόεδρος Αλμπασίρ ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις της πρόεδρου και μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε πρώτα με το σημείο 6, την πρώτη ανταλλαγή σύντομη ελπίζω απόψεων, επί της ετήσιας έκθεση για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2010. Η συγγετής του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό είναι η κυρία Ανδρικένε, αντιπρόεδρος της υποεπιτροπής μας και θα θυμάστε ότι ο είπα, η είπα, εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, υπέβαλε αυτή την έκθεση στην Ολομέλεια του Ιουνίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα πολύ συμμετείχατε στη συζήτηση που έγινε τότε που επικεντρώθηκε γύρω από τρία σημαντικά θέματα. Είχαμε την ετήσια έκθεση, την έκθεση για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ψηφίσματα για τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια που θέλουμε να αναθεωρηθεί είπατε εκπρόσωπος στην ομιλία της στην Ολομέλεια, είπε ότι είναι πρόθεσή της να αναθεωρήσει την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από φέτος. Οπότε, μέσω του εισηγητή της, η Υποεπιτροπή θα έχει μια ευκαιρία και μέσω της ετήσιας έκθεσης να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διαφωτίσει και την ύπατη εκπρόσωπο για το τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει αυτή η νέα στρατηγική. Αν ας ακούσουμε την εισηγητριά μας, την κυρία Αντρικένα. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, τα λιθονικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει τώρα να συντάσει την ετήσια έκθεση για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά από την παρουσίαση της υπάτης εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έκθεσης για την δράση της Ένωσης υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο. Η δική μας έκθεση θα περιλάβει ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο αφού θα αρχίσει από 1η Εβδόμου 2008 μέχρι τα τέλη του 2009, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Θα υπάρξει δυνατότητα να αναλυθεί η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, στα πλαίσια μιας δομημένης ανάλυσης που θα προσφέρει ένα εργαλείο όχι μόνο για τη διαμόρφωση της ε, ενωσιακής πολιτικής στον τομέα αυτό, αλλά θα προσφέρει και ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συντονιστούν οι πολιτικές στον χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε ποιο πλαίσιο λοιπόν θα συνταχθεί η έκθεση αυτή. Η περίοδος που θα καλύψει η ετήσια έκθεση συμπίπτει με την απρόσμενη τότε ε, δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Θυμίζω ότι 19 του 2001 άρχισε αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Είδαμε στην περίοδο αυτή και ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως της Κίνας, των Ινδιών και της Βραζιλίας που μπαίνουν πλέον στα, στις αποκλειστικές λέσχες δεν μπορούμε να μιλούμε όμως παρόλα αυτά για ε, καλό ιστορικό τους των ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ συχνά παραμελούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συζητήσεις με τις χώρες αυτές. Εκτός από τα οικονομικά πάντως και άλλα δημοσιονομικά προβλήματα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και την, ε, τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος που ίσως σας φανεί παράδοξο, αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μιλώ μόνο για τις πιο ευάλωτες ε, ομάδες πληθυσμού, όπως οι θαγενείς στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά η αλλαγή του κλίματος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το λοιπόν πολύ κρίσιμο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση όταν καλείται να μιλεί συστηματικά και διαρκώς για την ανάγκη βελτιώσεως των ανθρώπινων δικαιωμάτων με χώρε οι οποίε βρίσκονται εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενταχθούν σε όλους τους τομείς, να γίνει το mainstreaming δηλαδή, σε όλους τους τομείς ε, τη ε, της, ε, της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις με άλλες χώρες μέλη και εταίρους. Είναι σημαντικό λοιπόν στο πλαίσιο που σας περιγράφω να βάλω και την συνθήκη της Λισαβόνας η οποία, η άρχισε ε, να ισχύει ε, τρέχοντας το 2009 και η οποία ε, εισάγει πολλές καινοτομίες στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής με κύριο στόχο να ενισχυθεί η αξία των πολιτικών της Ένωσης και να τονιστούν οι αξίες, αξίες όπως δημοκρατία, αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Επίσης σε αυτά περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αρχές που θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αποτελέσουν την, τους πυλώνες του οποίους θα βασιστεί αυτή η εξωτερική δράση, τα θεμέλια. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να ε, συζητηθεί εδώ σε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση είναι η δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης με τα διάφορα συμπαροματούντα εξωτερικές ε, σχέσεις, ανθρωπιστική βοήθεια, διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις. Ο συντονισμός όλων αυτών των πολιτικών θα ανοίξει ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει να ακουστεί η φωνή της περισσότερο στις συζητήσεις με τους εταίρους της, με τις άλλες χώρες δηλαδή. Δεν θα υπησέλθω σήμερα σε λεπτομέρειες, διότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Αλλά όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά που λέω είναι σημαντικά. Και ο, η θέση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εμφανής. Σε αυτή την ετήσια έκθεση πρέπει να συζητήσουμε και τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρώτα-πρώτα βέβαια τις κατευθυντήριες γραμμές που είναι το βασικότερο εργαλείο που διαθέτουμε για την διαμόρφωση της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές που όπως λέω έχουν μεγάλη σημασία. Υπάρχει και το διεθνό, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το δεύτερο εργαλείο που έχουμε είναι ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις των χώρων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το τρίτο είναι το εργαλείο δημοκρατίας είναι η συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς. Στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και ούτω καθεξής. Και εκεί πρέπει να θέσουμε τα θέματα παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες. δεν, ναι, νομίζω ότι πρέπει να κατευθύνει τις σκέψεις μας αυτή η αρχή που στα αγγλικά λέγεται naming and shaming, αλλά παρόλα αυτά ορισμένα πράγματα πρέπει να καταγγέλλονται. Για παράδειγμα, η εκτέλεση θανατικών καταδικών πρέπει να ε, τονιστεί ιδιαίτερα στην έκθεση αυτή. Επίσης, η ε, ελευθερία θρησκευτική λατρείας, οι δραστηριότητες των ε, υπερμάχων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες. Βέβαια, ο κατάλογος αυτών των θεμάτων δεν είναι εξαντλητικός που σας αναφέρω και είμαι βεβαία ότι κατά την διάρκεια της συντάξεως της εκθέσεως θα έρθω και θα μου έρθουν και άλλες ιδέες άλλωστε και στις συζητήσεις με τους συναδέλφους μου και με τις ε, μη κρατικέ οργανώσεις επίσης και πολύ θα χαρώ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων μου σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ την φίλη κυρία Αντρικίανη. Καλά κάνατε και είπατε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τη στρατηγική αυτή. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αρχιτεκτονικής στη διεθνή κλίμακα. Πράγματι θα πρέπει να δώσουμε μια στρατηγική απάντηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να δούμε τι μορφή θα λάβει σήμερα αυτή η νέα στρατηγική. Ξέρετε ότι στην αρχή της εβδομάδας έγινε μια συζήτηση σχετικά με αυτή τη νέα στρατηγική ενόψη του φόρουμ με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και η κυρία Ντεκάιζερ προείδρευε μια ομάδα εργασίας σχετικά με τη στρατηγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Βελγική Προεδρία και η Κομισιόν είπαν ότι θα λάβουν υπόψη τους ό,τι υπόθηκε σε αυτό το φόρουμ. Και τώρα έχουμε την ε, ευκαιρία να τα ξαναπούμε με την έκθεση της κυρίας Αντρικάιν. Έχουμε ένα τέταρτο λοιπόν να ακούσουμε την, τις τοποθετήσεις σας. Θέλει κανείς να μιλήσει. Thank you. It's very difficult, of course. Δύσκολο να σχολιάσει κανείς το τεράστιο εύρος αυτής της ε, έκθεσης. Δεν έχω τίποτε νέο να προσθέσω στα όσα είπατε κυρία Ανδρικένε. Διαβάζοντας το πρώτο σχέδιο προμηνών, θυμάμαι ότι μου φάνηκε ότι η εισαγωγή της εκθέσεως ήταν πολύ καλή σε ό,τι αφορά την ε, μνήα της ανάγκης να υπάρξει καλύτερη συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζοντας όμως τα κεφάλαια, διαπίστωσα ότι αυτό δεν το πάντοτε σε όλα τα κεφάλαια, δηλαδή αναφέρω το παράδειγμα του follow-up που δίνουμε στις έκτακτες εκδόσεις της CIA με τις περίφημες εκείνες πτήσεις. Λέτε τώρα ότι στο πλαίσιο της εκθέσεως αυτής θα εξετάσετε και την οικονομική κρίση καθώς και τους αντικτύπους της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί ίσως μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη να δουλέψουμε και περισσότερο πάνω στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και στο τι σημαίνουν αυτά. Ίσως δεν τα παίρνουμε υπόψη στην έκθεση ακόμα όσο θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λόχ Μπίλερ. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κι άλλους. Ο αντιπρόεδρος μας. ο Αυτή η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και κοίταξα και τις προηγούμενες εκθέσεις, αλλά σε αυτή την έκθεση ειδικά είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αναλύουμε περισσότερο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Μιλάμε για στόχους πολύ συγκεκριμένους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ξεχνάμε να αναρωτηθούμε ποια είναι πραγματικά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σε αυτή την έκθεση ε, με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων. Έχω μία πρόταση, δεν ξέρω αν είναι εφικτή. Μία έκθεση αποτελεί κυρίως περιγραφή. Περιγράφονται δηλαδή διάφορες καταστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν σε μία τέτοιου είδους περιγραφή και σύνθεση να μην μιλήσουμε και για τις τάσεις Δηλαδή, ποιοι είναι οι τομεί εκείνοι όπου είχαμε μια χειροτέρευση, ποιοι εκείνοι που είχαμε μια σταθεροποίηση, ποιοι εκείνοι όπου παρατηρήσαμε βελτιώσει. Έτσι λοιπόν, συγκρίνοντας τις εκθέσεις χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε και τις τάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει το λόγο? Μία προσθήκη για τους ε, δύο συναδέλφους και θα ξαναδώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρό μας. Εμείς έχουμε ένα οριζόντιο ζήτημα, το συναντάμε παντού. Τι γίνεται με την συνοχή των διαφόρων δραστηριοτήτων μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να συναντήσουμε από την κυρία Γιάν που είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για τον ε, οργανισμό. Εμείς ε, μία φορά το χρόνο έχουμε μία έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και μια άλλη έκθεση σε εσωτερικό επίπεδο. Αυτά είναι τα μόνα πράγματα που κάνουμε και πολλές φορές δεν απολύγουν πουθενά αυτές οι εκθέσεις. Δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να εξετάζουμε αυτές τις εκθέσεις ταυτόχρονα θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και μια ταυτόχρονη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις δύο εκθέσεις. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από την κυρία Άστον και από την κυρία Ρέντινγκ να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση εάν θέλουν να ενοπίσουμε δηλαδή αυτές τις εκθέσεις και να έχουμε τέλος πάντων μια ουσιαστική συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ζάμπκε μας έκανε μια εξαιρετική πρόταση. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τάσεις. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κατάσταση των στρατευμένων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς αντιμετωπίζονται στις διάφορες χώρες και να δώσουμε διάφορα παραδείγματα. Κυρία Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ όλες και όλους τους ε, συναδέλφους Λόχμπιλερ, Ζέμκε και την Πρόεδρο για τα σχόλια και τις ιδέες που, συνέβαλαν, που συνεισέφεραν. Συγγνώμη. Τις δέχομαι. Η πρότασή σας να μιλήσουμε για τις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ένωσης και εντός και εκτός των συνόρων Αυτό μπορεί να συζητηθεί εκ παραλίλου στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα. Θα μας επιτρέψει έτσι να τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει δεκτό και από άλλους συναδελφούς, δεν ξέρω τώρα εάν ε, θα συμφωνήσουν. Δεν μπορούμε πάντως να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να... οι απαιτήσει να είναι ίδιες και για αυτούς που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσης και για αυτούς που βρίσκονται εκτός. Και ένα άλλο θέμα. πώς μπορεί να μετρηθεί μια κατάσταση ανθρώπινων δικαιωμάτων, στη βάση ποιων δικτών. Το Κοινοβούλιο κατά επανάληψη έχει ζητήσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο να προτείνουν τέτοια κριτήρια. Μέχρι τώρα αυτό δεν επιτεύχθη. Ελπίζω ότι με την έκθεση αυτή θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο εν προκειμένου. Πάντως παραμένω ανοιχτή στις ιδέες σας, στις ιδέες και στις προστάσεις σας και θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντάξω μια έκθεση που θα απηχεί όχι, βεβαίω, όχι βεβαίως μόνο τις δικές μου απόψεις και του κόμματός μου αλλά θα απηχεί τις απόψεις του Κοινοβουλίου για την κατάσταση ανά τον κόσμο. Ελπίζω να έχουμε και το χρονοδιάγραμμα σύντομα για την πρόοδο της εκθέσεως. Για τις προθεσμίες θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Δάμσκης. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις ιδέες της Προέδρου και της Αντιπροέδρου. Όντως πρέπει να αποκλείουμε κάθε ιδέα διπλών μέτρων και σταθμών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδίως όταν ε, πρόκειται, πρόκειται θέματα, όταν υπάρχουν μάλλον θέματα ε, επιθέσεων κατά του τύπου. Αν θέλουμε το ειδικό βάρος μας και η φήμη μας στα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι σεβαστά και καθαρά, πρέπει να αποφύγουμε κάθε ιδέα εφαρμογής διπλών ε, μέτρων και σταθμών ευχαριστώ κύριε Ντόμφκης Θα δούμε το χρονοδιάγραμμα. 30. Ε, με το χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί μία πρόταση. Θα το εξετάσουμε λοιπόν το θέμα στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο στην ε, υποεπιτροπή μας και 9 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια. Α, διορθώνεται η Πρόεδρος, το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο. Θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο λοιπόν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και στο εξωτερικό ταυτόχρονα στην Ολομέλεια και θα πρέπει στο μεταξύ να σκεφτούμε και σε ποιους θα δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ. Πρέπει να συνενώσουμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία για να έχουμε μια εκτενέστερη συζήτηση. Η συγγήτριά μας λοιπόν συμφωνεί για αυτό το σημείο ότι θα πρέπει να, να έχουμε συζήτηση για αυτό το θέμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ένα άλλο σημείο σχετικά με τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για την έκθεση της Αντιπροέδρου μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα συζητήσουμε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο σημείο 5 ανταλλαγή απόψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Νοτιοανατολική Ασία. Θα εξετάσουμε την κατάσταση τεσσάρων χωρών, του Βιετνάμ, της Καμπότζης, του Λάος και της Ταϊλάνδης. Έχουμε ελάχιστο χρόνο βέβαια για πάρα πολλές χώρες. Ίσως μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις χώρες γενικά, φυσικά είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά πρώτα γίνει μια γενική παρουσίαση και μετά να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους. Έχουμε προσώπους της κοινότητας Μπάτνα, που είναι μια θρησκευτική βιετναμική κοινότητα. Είστε εδώ, α, είστε εδώ στο βάθος της αίθουσας, καλωσορίσατε. πριν από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση σας ε, θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε πολλές φορές την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες. Κυρίως μετά από τις ε, συγκρούσεις και τα βία επεισόδια στην Ταϊλάνδη εξετάσαμε το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας στο Βιετνάμ, εξετάσαμε την κατάσταση των, προσφύγων, των Ιουγούρων προσφύγων, είναι μια κοινότητα που απειλείται ιδιαίτερα στην Κίνα, και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αργεί ιδιαίτερα στη λήψη των αποφάσεων. Και έχουμε βέβαια και την Καμπότζη. Τώρα, για το Βιετνάμ και για το Λάος έχουμε την μειονότητα Μπόγκ, η οποία εκδιώχθηκε βία προς το Λάος. Με μεγάλη χαρά Καλωσορίζω την ε, Σοφή ε, Ρίτσαρτσον. Την ε, συναντήσαμε στη Ουάσιγκτον όταν μια αντιπροσωπεία μας επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον. Η κυρία Ρίτσαρτσον είναι δικηγόρος του Human Rights Watch, του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καλώς όρισε Σοφή. Ελπίζουμε ότι με την παρουσίασή σου θα, έχουμε, θα διαμορφώσουμε μια σαφή ιδέα για την κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, 10 λεπτά λοιπόν Σοφή Ρίτσαρτσον. Ευχαριστώ την υποεπιτροπή σας Ευχαριστούμε την κυρία Χάουταλα για την πρόσκληση, αλλά και το Κοινοβούλιο γενικώ, γιατί εξακολουθεί να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την κατάσταση στις χώρες αυτές και χαίρομαι για το ψήφισμα που υιοθετήσατε για τη Βόρεια Κορέα. Πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω να, καλύψω τέσσερις ε, χώρες σε δέκα λεπτά. Ε, Στην Καμπότζη έχουμε πολλές παρενοχλήσεις, ε, βία, μεταχείριση εκτιβιστών, ε, κριτικές κυβέρνησης ε, κατά δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης, ε, παράνομες δικαστικές αποφάσεις, ε, ανεπαρκή προστασία των έτων άσυλο και τιμωρησία των αξιωματούχων των κυβερνήσεων που κατηγορούνται για καταχρήσεις. Θα επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί μου είπα να επικεντρωθώ σε θέματα της δικαιοσύνης. Η ΧΜΕΡΟΥΖ ε, ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε την, την απόλυση ενός ε, δικηγόρου τελευταία στιγμή όταν ζήτησε την αθώση ενός κατηγορούμενου. Σημαντικές κατηγορίες διαφθοράς επίσης κατά δικαστών που υπονομεύουν το δικαστήριο. Η παρέμβαση του Προέδρου στη, στο έργο της δικαιοσύνης είναι απαράδεκτη. Έτσι αποθαρρύνονται οι Καμποτζιανοί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι το διεθνές, η διεθνής αρρωγή θα βοηθήσει μόνο αν συνεχιστούν οι διεθνείς επικρίσεις κατά τις στάσεις της Καμπότζης, γιατί προς τι να δίνονται κονδύλια και επιχορηγήσει. αν δεν παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυ τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων. Έχουμε μετούντες άσυλο από Βιετνάμ, Κίνα, που πολλέ φορέ επαναπατρίζονται υποχρεωτικά, παρόλο που ε, αντιμετωπίζουν απειλέ ε, φυλακισμού και βασανιστήριων. Μάλιστα, το Δεκέμβριο του 2009 είχαμε τέτοια παραδείγματα ε, υποχρεωτική επιστροφής χωρίς να, να εξεταστούν καν ε, δεόντω οι φάκελοι του παραβιάζονταν, παραβιάζονται σημαντικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Παρόλο που τέτοιες ε, διεθνείς συμβάσει έχει επικυρώσει η Καμπότζη. Μάλιστα το Δεκέμβριο του 2009 υιοθετήθηκε ένα διάταγμα από την Καμπότζη που κατά τη γνώμη μου δεν συμπεριλαμβάνει τον ορισμό του πρόσφυγα από διεθνείς συμβάσεις, ούτε εξασφαλίζει προστασία για τους πρόσφυγες. Άλλωστε δεν τηρεί και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή η Καμπότζη. Και μάλιστα δεν θα πρέπει ο προσδιορισμός ε, τη... του ορισμός του πρόσφυγα να απαφίεται στην διακριτική ευχαίρεια της καμποζέινης κυβέρνησης. Και μάλιστα θα πρέπει ε, και η αρμόδια οργάνωση του ΟΗΕ να εξασφαλίσει την προστασία των ε, προσφύγων. Και με δύο λόγια να μιλήσω για το Λάος. Θα σας δώσω ακόμη λίγα λεπτά, γιατί πραγματικά είναι αδύνατο να καλύψετε τόσες χώρες σε τόσο λίγο χρόνο. Ευχαριστώ που σέβεστε και τα δικά μου ανθρώπινα δικαιώματα. Γενικώ για το Λάος η κυβέρνηση υποβάλλει σημαντικού περιορισμού σε θέματα συγκέντρωση ε, του συνεταιρίζεστε και τη έκφραση πολιτικών δικαιωμάτων. Μου είπατε σήμερα το πρωί να επικεντρωθώ στο θέμα του, των πρόσφυγων ΜΟΝΚ και την, ε, τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό του στην Ταϊλάνδη το Δεκέμβριο του 2009. Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικέ ομάδες. 150 ε, ΜΟΝΚ που αναφέρονται ως η ομάδα των Ρονκάη, είναι άνθρωποι που έχουν προσφορές ε, από Καναδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία για φιλοξενία εκεί. 4.500 μόγκ βρίσκονται σε ένα καταβλισμό προσφύγων. Και 800 από αυτούς ε, έχουν προβλήματα και απειλές, αντιμετωπίζουν απειλές στην Ταϊλάνδη. Επίσης, και κάποιοι από την ομάδα Νονκάι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Βέβαια, έχει καταδικαστεί επίσημα η Ταϊλάνδη για την ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη χρήση βίας και απειλή χρήσης βίας προκειμένου να ξαναγκαστούν οι μόγκοι να φύγουν από τον καταβλισμό προσφύγων, ιδιαίτερη ομάδα Νονκάι, και να ε, ξαναγυρίσουν στο Λάος και μάλιστα είχαμε υποχρεωτικές, ε, υποχρε... υποχρεωτικούς ε, εκτοπισμούς σε δύο πόλεις που δυστυχώς δεν τις έχω προφέρει καλά. Μάλιστα στους καταβλισμούς αυτούς δεν υπάρχει καν ηλεκτρισμός, ε, αποχετευτικό σύστημα, δεν υπάρχει σωστή διατροφή, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παιδεία και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες για παρενόχληση από την κυβέρνηση και υπάρχουν και προβλήματα με τη διανομή των γεών γύρω και με τη γεωργία στην γύρω περιοχή από τον καταβλισμό. Δυστυχώς οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από την κυβέρνηση είναι αναξιόπιστες για να μην πω τίποτα χειρότερο και είναι πολύ δύσκολη η παρακολούθηση κατάσταση. κατάστασης. Μάλιστα η κυβέρνηση επέβαλε μια απαγόρευση κυκλοφορίας για ορισμένα μέλη της ε, ομάδας απαγορεύοντας την επιστροφή του στην Ταϊλάνδη. Και μάλιστα η κυβέρνηση του Λάους είπε ότι θα εκδώσει ταυτότητες προκειμένου να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα οι πρόσφυγες, αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις, ούτε η υπόσχεση που δόθηκε στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να επιτρέψει πρόσβαση της διεθνούς κοινότητας στους καταβλισμούς και να επιτρέψει ορισμένους να εγκατασταθούν σε περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση από άλλες χώρες. Είχαμε το πρωί αρκετά λεπτομεριακή συζήτηση με εκπροσώπους της ε, γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκαν το Λάος, προσπάθησαν να επισκεφθούν τους καταβλισμούς προσφύγων, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν ε, ε, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη που ζήτησαν. Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης και για τους ξένους δημοσιογράφους και για τους διεθνούς παρατηρητές. Βέβαια, δύο από την ομάδα Νονκάη κατάφεραν να, να διαφύγουν και να επιστρέψουν στην Ταϊλάνδη. Προς το παρόν ε, την χάνουν τους δύο προστασίες, αλλά το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Πάντως, ε, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ε, δεν δίνει εξόδους άδειας για τους Μόγκ που έρχονται από το Λάος. Εμείς συστήσαμε στην κυβέρνηση του Λάος να επιτρέψει η ελευθερία έκφρασης και διακίνησης του ΣΜΟΝΚ, ώστε να μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα στο Λάος και να επιστρέψουν στις χώρες που τους προσκαλούν και επίσης να εξασφαλίσουν πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων του ΟΗΕ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των προσφύγων, να αποφύγουν παρενοχλήσεις ιδιαίτερα για την ομάδα Νονκάη να άρουν την απαγόρευση κυκλοφορίας εντός του καταβλισμού και να επιτρέψει την ύπατη αρμοστία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να επισκεφθεί τη, τους καταβλισμούς. Επίσης, και η κυβέρνηση του Λάου θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα της καταδίωξης και της διακριτικής μεταχείρισης κατά τον ΜΟΝΚ. Προτείναμε στην κυβέρνηση Ταϊλάνδης ε, να εκδώσει τις άδειες εξόδου, όσοι έχουν ε, προσφορές επανεγκατάστασης να μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. Πολύ ευχαρίστως ε, να συζητήσουμε το θέμα της παλινδρόμησης που έκανε η Ταϊλάνδη ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων, που δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στο Λάος αλλά και σε άλλες χώρες. Τώρα για την Ταϊλάνδη. Μας ε, ανησυχεί ιδιαίτερα η τρίμηνη παράταση της, ε, του διατάγματος εκτάκτου ανάγκης ε, για την Παγκό και 18 άλλες ε, επαρχίες μέχρι ότου επιστρέψει η κατάσταση σε μία ομαλότητα. Βέβαια το διάταγμα αυτό αναστέλει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται και από το Ταϊλανδέζικο Σύνταγμα και νόμο καθώς και από το Διεθνές Δίκαιο. Δεν δικαιολογείται η κατάσταση στη Ταϊλάνδη για την αναστολή τόσο σημαντικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλιστα, μια, ένα τέτοιο δικαίωμα είναι η παράταση της φυλάκισης ανθρώπων που δεν έχουν καν κατηγορηθεί. Δεν δίνονται εχέγγυα κατά των καταχρήσεων και της κακομεταχείρισης αυτό που βρίσκονται σε κράτηση. Συνοπτικές διαδικασίες ε, για εγκλήματα που εμπίπτουν στο διάταγμα, λογοκρισία και ούτω καθεξής. Επίσης ε, ασκήθηκε βία και από κυβερνητικές και από αστυνομικές δυνάμεις κατά των, ε, της ομάδας των κόκκινων υποκαμίσεων. Οι δημοσιογράφοι ε, υπέσαν απειλές. Σοφία, μιλάς πολύ, πολύ γρήγορα. Θα μπορούσες να μιλήσεις λίγο πιο αργά. Επίσης έχουμε λάβει ανησυχητικές εκθέσεις ότι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και νοσηλευτικό προσωπικό υποχρεώθηκαν να αναφερθούν στο CRS e όταν είπαν ότι ήταν αυτό τις μάρτυρες καταχρήσεων εκ μέρους των κυβερνητικών και αστυνομικών δυνάμεων. έχουν φυλακιστεί ε, ακτιβιστές και άνθρωποι που έκαναν διαμαρτυρίες. Η, η κυβέρνηση δεν δίνει ακριβή στοιχεία για τους κρατούμενους, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε σε ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα η κυβέρνηση δεν δίνει πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό φυλακισμένων ε, με βάση το έκτακτο προεδρικό διάταγμα της 7ης Απριλίου, ούτε δόθηκαν τα ονόματα, το καθεστώς και τα, το μέρος φυλάκισης αυτών των ε, ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση εκεί τα μέλη της οικογένειάς τους ή δικηγόρη τους. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα πάνελ για να διερευνηθούν οι καταχρήσεις ε, που έχουν λάβει χώρα από τον Απρίλιο με το έκτακτο προεδρικό διάταγμα και έχουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, δικηγόρων που υπέσαν απειλές. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κολυσιεργία που διαπιστώνεται σε ό,τι αφορά τη σύσταση αυτού του πάνελ. Και δεν ξέρουμε αν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει καταρχήν να αρθούν ε, οι περιορισμοί στα μέσα μαζική ενημέρωση και να ανασταλεί το έκτακτο προεδρικό διάταγμα, ώστε οι διώξει να γίνονται με ισότιμο τρόπο και όχι με διακριτική μεταχείριση. Το έκτακτο αυτό διάταγμα ε, ισχύει στη Νότια Ταϊλάνδη από το 2005 και όλοι οι περιορισμοί που ανέφερα είναι ουσιαστικά καθημερινότητα στην Νότια Ταϊλάνδη. Και η δικαιολόγηση της κυβέρνησης είναι ότι προσπαθεί να περιορίσει τους αντάρτες, αλλά η Human Rights Watch έχει, ε, επισημάνει σημαντικές παρενοχλήσεις, βασανιστήρια, εξαφανίσεις ε, που διαπράττονται από ε, δυνάμεις ασφαλείας κατά των κρατουμένων. Και έχουμε συγκεκριμένες περιστάσεις και συγκεκριμένες παραβιάσεις κατά ακτιβιστών. Και μάλιστα οι στρατιωτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν βασανιστήρια. Αυτές οι πόνες τουλάχιστον υπάρχουν κατά των κρατουμένων. Και μάλιστα πρώτη, ε, έχουμε την πρώτη γνωστή περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της κράτησης. Ε, βασανίστηκε μέχρι θανάτου σε ένα στρατόπεδο και μάλιστα χάρη στην ε, διεθνή πίεση ο επικεφαλής στρατηγός δήλωσε ότι οποιοδήποτε ε, υπέτειος θα τιμωρηθεί. Βέβαια δεν υπήρξε καμία ούτε δίκη ούτε κατηγορία καταστρατητικού για την περίπτωση του Μαριάπαρ, ούτε και για καμία άλλη κατηγορία κατάχρησης από πλευράς ε, στρατιωτικών κατά των ε, φυλακισμένων στην νότια επαρχία της Ταϊλάνδης. Ο μόνος τρόπος για να αρχίσει μια επανασυμφιλίωση στη νότια Ταϊλάνδη είναι να σταματήσει ο κύκλος της ατιμορρησίας. Θα πρέπει και τα μέλη της κυβέρνησης να προσάγονται στα δικαστήρια και οι αντάρτες επίσης. Δεν μπορούν να υλοσκοτώνονται η μέρμα με τους δε και να χαίρουν τις ατιμορρησίας. Είναι μια ανοιχτή πληγή αυτή η περίπτωση της Νότιας ε, Ταϊλάνδης και θα πρέπει η κυβέρνηση να τη διορθώσει. Τώρα για τους ε, μετανάστες που συνεισφέρουν το 6% του ΑΕΠ στην ε, Ταϊλάνδη, η Human Rights Watch έχει συντάξει έκθεση για τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων σε βάρος των 800 περίπου χιλιάδων ε, μεταναστών που έρχονται από το Λάος και από άλλες χώρες οι οποίοι έχουν περιγράψει ξυλοδαρμούς και άλλα βασανιστήρια ακόμα και ε, σεξουαλικές καταχρήσεις κλπ και ε, εν τέλει απελάσεις. Την 1η Μαρτίου ε, απέτησαν οι αρχές στην Ταϊλάνδη όλου, από όλους τους μετανάστες να καταχωριστούν ή να σηκωθούν να φύγουν. Εμείς συστήσαμε οι απελάσεις να σταματήσουν και όσοι έχουν σοβαρούς λόγους να ζητήσουν άσυλο να ε, τους επιτραπεί να απευθυνθούν στις αρμόδιες οργανώσεις. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης θα πρέπει να συνεργαστεί με τον εκπρόσωπο των Εθνών για να κάνει τις απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία. Τώρα που η Ταϊλάνδη είναι και μέλος της, ε, ε, του Συμβουλίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων έχουμε και περισσότερες απαιτήσει από αυτούς για τη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς διατάξεις των, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, Βιετνάμ. Προχωρώντας προς το επόμενο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, η κυβέρνηση ε, προβαίνει σε καταπιεστικές ε, δραστηριότητες για να ενισχύσει έτσι το κύρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρενοχλώντας ε, τους διαφόρους οι οποίοι τάσσονται υπέρ δημοκρατικών ανοιγμάτων. Έχουν Παρενοχλούνται επίσης ε, ε, διάφοροι που έχουν ε, blogs στο διαδίκτυο και άλλα σχετικά. Η κυβέρνηση στο Βιετνάμ εξακολουθεί να απαγορεύει τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα και άλλες οργανώσεις, καθώς και πολιτικά κόμματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα βαριάς πολιτικής καταπίεσης μπαίνουν στη φυλακή όσοι τολμούν να αμφισβητήσουν το κύρος της κυβερνητικής εξουσίας. Η χρήση αστυνομική βίας είναι διαρκής και κυρίως σε ό,τι αφορά τις ανακρίσεις πολιτικών και θρησκευτικών κρατουμένων οι οποίοι ε, στερούνται των επισκέψεων των μελών της οικογένειάς τους, ε, συχνά ε, σε, βάζουν σε δίκες χωρίς συνήγορο και καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης. Ε, με κατηγορίες όπως αντικυβερνητική προπαγάνδα ή ότι καταχρώνται, λέει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ, των δημοκρατικών ελευθεριών. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ εξακολουθεί να επιμένει ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση δηλαδή να ρυθμίσει το τι θα πιστεύει ο καθένας για την, ε, θρησκευτικές του πεπιθήσεις δηλαδή. Υπάρχουν και προβλήματα ε, κατοχής γης. Η συμμετοχή σε μη καταχωρημένες θρησκευτικές οργανώσεις, όσοι δηλαδή ε, κατηγορούνται γι' αυτό, παρενοχλούνται και ε, κρατούνται κατοίκων. Και πέρσι μάλιστα εκτοπίστηκαν νεαροί μοναχοί και μοναχές από βουδιστικό μοναστήρι. Έχουν γίνει κατασχέσεις εκκλησιαστικών περιουσιών σε ορισμένες πόλεις και μάλιστα και ορισμένοι που διαμαρτυρήθηκαν τελικά ε, φωνεύθηκαν. Θα θέσω υπόψη σας ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις βουδιστών μοναχών Μαχά και Μάιτι Ντόγκ. Το 2005 και 2006 συνελήφθησαν 12 μοναχοί, βουδιστές μοναχοί, επειδή παρενόχλησαν τη δημόσια τάξη, διαμαρτυρώμενοι κατά της ε, κρατήσεως των θρησκευτικών ηγετών τους. Βουδιστές ΟΑΧΑ έχουν προχωρήσει σε απεργίες πείνας και σε αυτοπυρπολήσεις. Ένας από αυτούς επέζησε, ο άλλος απεβίωσε. Οι αρχές χρησιμοποιούσαν βία για να διαλύσουν τις ε, εκδηλώσεις που έγιναν στις των προσώπων, στην κηδεία ε, του προσώπου αυτού. Θα γνωρίζετε την περίπτωση του πατρός Win Βαν Λί που φυλακίστηκε για πολιτικές πεπιθήσεις παραπάνω από 15 χρόνια τώρα από το 1977 και πρόσφατα καταδικάστηκε το 2007 πάλι σε 8 χρόνια φυλακή για αντικυβερνητική προπαγάνδα. Τον Μάρτιο 2010 απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές για ε, λόγου υγεία, αλλά με τον όρο ότι θα επιστρέψει στις φυλακέ μόλις βελτιωθεί η υγεία του. Υπάρχει και στο διαδίκτυο ε, τεκμηρίωση για ευρύτατη χρήση βασανιστήριων. Ο πατέρας Λί θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινή του και είναι απόλυτα απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει το θέμα του ε, πατρός αυτού για να γλιτώσει ο άνθρωπος όχι μόνο τη φυλακή αλλά και τα παραπέρα βασανιστήρια. Μερικές συστάσεις για το Βιετνάμ. Θα θέλαμε να δούμε ε, ενεργό υποστήριξη των οπαδών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και ε, να σταματήσουν ε, δραστηριότητες της κυβέρνησης όπως παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων εκείνων που τάσσονται υπέρ των δημοκρατικών ελευθεριών. αυτά τα θέματα δεν μπορούν να περιοριστούν μοναχά σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όλοι οι ευρωβουλευτέ θα πρέπει να θέτουν τα θέματα αυτά σε όλες τις ε, συζητήσει με την κυβέρνηση του Βιετνάμ η οποία παραβιάζει όλες τις γνωστές συνταγματικές ελευθερίες. Πρέπει να τροποποιηθεί επίσης ο ποινικό νόμος στο Βιετνάμ και κυρίως η ε, πολύ ασαφείς διατάξεις του για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Σοβαρές, σοβαροί περιορισμοί στην χρήση του διαδικτύου και επίσης να ανοιχτεί η δυνατότητα για ανεξάρτητες ε, οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων να επισκέπτονται το Βιετνάμ και να επιζητούν ε, επαφές με πρόσωπα τα οποία έχουν Ευχαριστώ πολύ. Μας είπατε πάρα πολλά, πολλές πληροφορίες σε πολύ σύντομο διάστημα. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τους ε, πρέσβεις αυτών των χωρών, να καλωσορίσω και τον πρέσβη της Ταϊλάνδης. Είχαμε χθες την ευκαιρία να εξετάσουμε χθες τέτα την κατάσταση στη χώρα σας. Συζητήσαμε για την ασφάλεια, αλλά και το θέμα των ελευθεριών. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Υποεπιτροπής, κυρίες και κύριοι. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την Υποεπιτροπή σας για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ταϊλάνδη. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ταϊλάνδη και τη δηλώσει τη ΣΥΠΑ της εκπροσώπου για την Βαρόνι Άστον είναι ε, χαρακτηριστικά της επικοδομητικής τάσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ταϊλάνδη. Τα τελευταία χρόνια η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ταϊλάνδη υπέστησαν φοβέρε δοκιμασίε. Η κυβέρνηση από τη μια ε, θα πρέπει να τηρήσει και να σεβαστεί τα δικαιώματα των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να προστατεύσει και το κράτος δικαίου όταν απειλείται η δημόσια ασφάλεια. Και οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου είναι ε, λυπηρή. Βέβαια η κατάσταση έχει επανέλθει στην σε μια ομαλότητα, παρόλο που σε ορισμένε περιοχέ και επαρχίε χρειάζονται έκτακτα μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη τη βία. Έχω ετοιμάσει ήδη μια δήλωση, αλλά μια και δεν έχω χρόνο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο σημεία της. Από την αρχή ήδη η κυβερνητική προσέγγιση ε, απέναντι στους διαδηλωτές ήταν ε, να αποφύγει οποιαδήποτε αντιπαράθεση, να μην χρησιμοποιήσει βία και να επιτρέψει όλες τις πλευρές να εξασκήσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους με βάση το κράτος δικαίου και το Ταϊλανδέζικο Σύνταγμα. Όταν οι διαδηλωτές ε, το Μάρτιο του 2010 ξεκίνησαν οι ειρηνικές διαδηλώσεις, ζήτησαν άμεση διάλυση της Βουλής. Μετά τις 10 Απριλίου κατέστησα αφές ότι οι διαδηλώσεις αυτές πια δεν ήταν ειρηνικές, γιατί μία ομάδα χρησιμοποίησε όπλα κατά ε, αξιωματικών ασφαλείας και κατά αθών. Ε, χρειάστηκε λοιπόν κάποια μέτρα για να επανέλθουμε στη, στο κράτος δικαίου και να αποκατασταθεί ομαλότητα στην καθημερινότητα της α, νότιας επαρχίας. Με βάση το δικό χάρτη που συστάθηκε, ο Πρωθυπουργό πρότεινε τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης εξατιστικής επιτροπής για να εξηχνιαστεί η, να εξηχνιαστούν τα εγκλήματα του Απριλίου και μάλιστα ένας σημαντικός δικηγόρος και πρώην εισαγγελέα διορίστηκε πρόεδρος αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής που ήδη έχει ξεκινήσει την ερευνητική διαδικασία με συναντήσεις ηγετών των διαδηλωτών για να ακούσουν και οι δικές τους απόψεις. Επίσης θα γίνουν ακροάσεις με συμμετοχή ψυχιάτρων, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, κτλ. Μάλιστα, ο, ο πρόεδρος της εξεταστικής αυτής επιτροπής διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν οι αρχές αμεροληψίας, ειλικρινίας εντιμότητας, ακαιρεότητας και η εντολή της εξεταστικής αυτής επιτροπής θα προσπαθήσει να επουλώσει τα τραύματα και να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Η εντολή έχει διετή διάρκεια, θα ενημερώνουν τακτικά το κοινό ανάλογα με τα πορίσματα που θα συγκεντρώνει και τα τεκμήρια που θα συγκεντρώνει η Επιτροπή και μάλιστα και τα τοπικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ε, μπορούν να συνεργαστούν με την εξεταστική αυτή επιτροπή και να υποβάλουν ε, και στοιχεία. Θεωρούμε ότι η διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων ίσως ε, απαιτήσει την συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες και μάλιστα ίσως προσφύγουμε και στου εμπειρογνώμονε των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ανάμειξη του ΟΗΕ κατά ανάγκη στο έργο της εξεταστική αυτής επιτροπής. Ε, παράλληλα, η, Διεθνής, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η, Διεθνής, ε, και η Εθνική Επιτροπή Πάταξης Διαφθορά διενεργούν ανεξάρτητες έρευνες ε, από πλευρά του. Και μάλιστα η κυβέρνηση είπε ότι η, θα συνεργαστεί πλήρω με τι επιτροπές αυτές και θα αναλάβει τις ευθύνες των δράσεών της. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες για την ε, παράταση του έκτακτου διατάγματος, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της καταστρατήγης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια το έκτακτο διάταγμα δεν είναι κάτι άγνωστο ακόμη και για δημοκρατικές χώρες. Δεδομένης της κατάστασης που δημιουργήθηκε η χρήση του έκτακτου διατάγματος είναι απαραίτητη προς το παρόν. Αλλά θα περιορίσετε σε συγκεκριμένου τομεί. Τον Ιούνιο, μάλιστα, η Ταϊλανδέζικη κυβέρνηση ήρε την εφαρμογή του διατάγματος σε πέντε από τις 24 επαρχίες και έδωσε ε, διασφαλίσεις ότι το διάταγμα θα σταματήσει να, λειτουργεί, να ισχύει εφόσον πληρώσει την, ε, τον προορισμό του που είναι η εξασφάλιση προστασίας των πολιτών της Ταϊλάνδη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την πολιτική της Ταϊλάνδη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Πρέσβε, παρακαλώ μην διαβάζετε την έκθεσή σας. Ε, μπορείτε να μας τα πείτε συνοπτικά γιατί δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Έχουμε και του ομολόγου σα από άλλε χώρε. Παρακαλώ κάντε μα μια σύνοψη της ε, έκθεσής σας, γιατί τους ή άλλους ε, γραπτός θα την έχουμε και θα την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά, αλλά δεν χρειάζεται να μας τη διαβάσετε ε, διεξοδικά. Ήδη έχω περάσει το πεντάλεπτο, οπότε μπορώ να σταματήσω και τώρα. Θα έχω την ευκαιρία στη συζήτηση να συμμετέχω. Είστε πολύ γενναιόδωρος και το εκτιμώ ιδιαίτερος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τη δήλωσή σας. Θα επανέλθουμε σίγουρα στη συζήτηση στα θέματα αυτά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φαν Τι Μαν και τον κύριο Βου Τουαν Χάι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Έχετε κι εσείς πέντε λεπτά. Um, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, η κυβέρνηση του Βιετνάμ υποστηρίζει τα πορίσματα της πρόσφατης έκθεσης της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Βιετνάμ στη διάρκεια του 2010. Καμιά φορά διαφορές απόψεων που βασίζονται σε διαφορετική πληροφόρηση παραμένουν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, ε, Εθνικής Συνέλευσης του Βιετνάμ. Στο πνεύμα αυτό μέσα σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που μας επιτρέπει να θέσουμε υπόψη των μελών της υποεπιτροπής σας από πρώτο χέρι πληροφορίες για το Βιετνάμ. Θα σας αναφέρω ορισμένα από τα επιτεύγματα των τελευταίων μηνών του Βιετνάμ. Παρόλο που αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, η οικονομία του Βιετνάμ συνεχίζει την ανάκαμψή της. 5,8% είναι ο ρυθμός ανάπτυξης στους τελευταίους ε, μήνες και ε, για το πρώτο εξάμεινο του 2010 έχουμε φτάσει στο 6,5% παραπάνω από 300.000 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν και στη συνέλευσή μας έχουν ε, ψηφιστεί 20 νομοθετήματα για παράδειγμα για την προστασία των αναπήρων, ε, των αναπήρων παιδιών και διάφορα άλλοι νόμοι. Στον τομέα των θρησκειών διάφορες δραστηριότητες αναλαμβάνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα η Καθολική Εκκλησία ε, διοργανώνει εκδηλώσεις με συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ε, ε, πιστών και με συμμετοχή και εκπροσώπων του Βατικανού. Το ίδιο για τους βουδιστές με διάφορες εκδηλώσεις στο Ανόη θα γίνει φέτος, τον Νοέμβριο δηλαδή, ε, το έκτο συμβούλιο των ε, βουδιστών Σανχά. Οργανώθηκε και με παραπάνω από 3.000 συμμετοχές ε, μεγάλη, μεγάλη ε, διάσκεψη οργανώσεων στο Βιετνάμ. Λυπούμεθα ωστόσο που οι πληροφορίες που σας παρέχονται σχετικά με την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα από ορισμένα άτομα ή οργανώσεις που είναι πάντοτε ανακριβή ή είναι κατασκευασμένα με κακές προθέσεις, με πρόθεση μάλλον να βλάψουν το Βιετνάμ. Ανακριβείς πληροφορίες που λένε ότι το Βιετνάμ δεν έχει ανταποκριθεί σε πολλές από τις συστάσεις που έγιναν από τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Το ε, ε Βιετνάμ πέρσι επενέθηκε για, τις, για τα επιτέματά του από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Λάβαμε 123 συστάσεις από τις οποίες έχουμε υλοποιήσει σχεδόν τις 100 και πάντως πάνω από το 75% είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέλη των ΗΕ, ενώ ορισμένε χώρες μεταξύ αυτών και ε, μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υλοποιήσει μέχρι και 40% των ε, σχετικών συστάσεων. Έχουμε λοιπόν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές. Έχουμε προσκαλέσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να επισκεφθούν το Βιετνάμ και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και το την εδώ την ε, ε, εβδομάδα, ειδικό απεσταλμένο για τα θέματα των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Συνεχίζουμε τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πολλές χώρες και με ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένε Πολιτείες, την Ελβετία και την Ορβηγία. Δεύτερο, η ελευθεροτυπία, η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτά είναι εγγυημένα και, στον, ε, και στους νόμους αλλά και στην πράξη στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι πραγματική δύναμη για την εφαρμογή των ε, διατάξεων αυτών και ιδίως όσων αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Βιετνάμ, όπως λέτε και στην εκθεσή σας, ε, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές. Είναι τέτοια μεγάλη ανάπτυξη του τύπου και του ίντερνετ που δεν μπορεί να πει κανεί πλέον ότι υπάρχει ε, σφιχτός έλεγχος των ε, μέσων αυτών στην, στο Βιετνάμ. Διότι αν υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί που ε, λένε ορισμένοι, δεν ε, θα είχαμε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Εμείς έχουμε 25.000 τόπους λατρείας στο Βιετνάμ. Τον Μάιο του 2009, όταν ο κύριος Μάικλ Λιούις, πρόεδρος της... Ε, είπε, τότε ότι σημειώνονται σημαντικές πρόοδοι στην άνοιξη στο Βιετνάμ με φροντίδα των τόπων λατρείας και των σχετικών θεσμών. Σας παρακαλώ κυρία, Πρέσβη, κυρία μία φράση και τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Οι πληροφορίες που σας δίνονται λοιπόν δεν είναι ακριβείς η σχέση μεταξύ του Βιετνάμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται θετικά. Ελπίζω λοιπόν ότι ο διαρκής διάλογος και οι ανταλλαγές απόψεων για ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνεχιστεί για να αποφευθούν οποιασδήποτε παρανοήσεις. Ναι, Εάν έχουμε λανθασμένες ε, πληροφορίες, ελπίζω ε, ότι θα μπορέσετε ε, να τις ανατρέψετε δημόσια. Γιατί όντως έχουμε λάβει πολύ ανησυχητικές πληροφορίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα σας. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά με χαρά μου προσκαλώ τώρα τον πρέσβη της Καμπότζης, κ. Νόν Ξακάλ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τα μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη. Η Καμπότζη είναι μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση το Σύνταγμα του 1996, το οποίο αναγνωρίζει την ελευθερία έκφρασης και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα. Από το 1993 η Καμπότζη έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ε, χίλιες περίπου ε, οργανώσεις ε, κοινωνίας των πολιτών και ελεύθερα συνδικάτα καθώς και ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης δραστηριοποιούνται στην Καμπότζη ενώ έχουμε το NDDI, AOI και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις καθώς και εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ. Σέβεται την ελευθερία έκφρασης, κυκλοφορούν πολλές ε, εφημερίδες, έχουμε 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς και 8 τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν αρκούν όλα αυτά. Υπάρχει πρόσβαση στο CNN και σε πολλά διεθνή δίκτυα και σταθμούς στην Καμπότζη. Σε ό,τι αφορά τις ε, δικαστικές αποφάσεις, ε, σε ό,τι αφορά κάποιες δυσφημίσεις και παραβιάσεις δικαίου, Έχουμε το άρθρο 61, 62 και 63 και σας παραπέμπω εκεί. Σε οποιαδήποτε δημοκρατική κοινωνία είναι σημαντικός ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Και φυσικά ε, ο σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Η ελευθερία έκφρασης δεν είναι απόλυτη και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται διακριτικά. Δεν θα πρέπει να γίνονται εκστρατείε παραπληροφόρησης και δυσφήμισης της καμποτζιανής κυβέρνησης. Και η ελευθερία έκφρασης ε, υπάγεται στην συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των γεών. Έχουμε σχετική νομοθεσία που αναγνωρίζει την, ε, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας της γης και εξασφαλίζει το δικαίωμα κυριότητας της γης η Εθνική Αρχή για, την, για το διακανονισμό διαφορών με τη γη, με, για τη γη συστήθηκε το 2006 και μάλιστα η καμποζιανή κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια πολιτική παραχώρησης ε, γεωργικών γεών σε ακτήμονες και σε φτωχούς και έχουμε παραχωρήσει αυτόν τον τρόπο πάνω από, το, από 4.000 εκτάρια στην νότια ε, επαρχία, αλλά και σε άλλες επαρχίες της χώρας. Στην Καμπότζη έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν παράνομα τα πεζοδρόμια και ε, είναι πλανόδιοι πολιτές ή επίσης ε, κάνουν καταλήψεις σε δημόσια κτίρια. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια κατάσταση χωρίς να προ... υιοθετούμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα. Τον Ιούνιο, ο ειδικό απεσταλμένος ε, στο ΟΗΕ για την Καμπότζη πραγματοποίησε δεκαήμερη επίσκεψη στην Καμπότζη. Στη διάρκεια της επίσκεψης αυτής συναντήθηκε με πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμανς, για να μας ενημερώσει για τα βασικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά αποστολές παρατήρησης ε, στις τέσσερις αυτές χώρες. Κύριε Τίμανς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την κατάσταση γενικώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Ασία, όπως την παρατηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τις χώρες, αυτές τις τέσσερις που εξετάζεται. Γενικώ πάντως θα έλεγα ότι έχουμε πολλές διμερείς δομές με πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίως το Βιετνάμ, την Καμπότζη και το Λάος. Και εκεί στις διμερείς αυτές επαφές εξετάζουμε τακτικά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη ότι πρόσφατα συστήθηκε η διακυβερνητική οργάνωση ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λειτουργεί πλέον πλήρως. Πρόσφατα συνεδρίασε στο Βιετνάμ υπό Βιετναμική Προεδρία προκειμένου να εγκρίνει το πενταετές πρόγραμμα εργασίας και εμείς ε, είχαμε επαφή με το γραμματέα της ΑΣΕΑΝ προκειμένου να βρούμε τρόπους ε, για να υποστηρίξουμε αυτή την ε, διακυβερνητική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΑΣΕΑΝ. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη είναι άκρος σημαντική. Γενικώ πάντως διαπιστώνουμε ότι σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Πιο διεξοδικά μας τα ανέφερε στην έκθεσή της η Σόφη Ρίτσαρτσον. Υπάρχουν προβλήματα μειονοτήτων, σε όλες τις χώρες, τα θέματα μετανάστευσης και προσφύγων επίσης, το θέμα του λαθρεμπορίου είναι σημαντικό ζήτημα και αφορά τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών και εμπορίου ανθρωπίνων όντων. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί και του δικαιώματο ελευθερία έκφραση και των δικαιωμάτων των μέσων μαζική ενημέρωση. Βέβαια, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν προβλήματα με την ελευθερία έκφρασης αλλά και εδώ η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες οπότε η ανάλυση θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση. Υπάρχουν προβλήματα και με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας και της υγείας. Δυστυχώς ε, υστερούν ε, αυτή η τομή σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες. Και υπάρχουν κάποια γενικά προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας αυτές. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη όπως θα έπρεπε κανονικά. Και δεν πληρούνται και τα εχέγγυα της ε, δίκαιης δίκης σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα προσαγωγές ε, στη δικαιοσύνη ακτιβιστών ή αντιφρονούντων. Γενικώ δεν υπάρχουν χέγγια δικαιοσύνης ε, όσων πέφτουν στα χέρια του δικαστικού συστήματος στις χώρες αυτές. Και σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, γιατί ασκούνται πιέσεις στην κοινωνία των πολιτών. Και λυπούμαστε ειλικρινά που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών δεν λειτουργούν τόσο ελεύθερα όσο θα έπρεπε. Και εμείς υποβάλλουμε κλίσεις στις χώρες αυτές, ώστε να υιοθετήσουν μια νοοτροπία που θα επιτρέπει τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εγγύσεις για την αηφόρα ανάπτυξη αυτών των χωρών και από οικονομική και από πολιτική άποψη. Υπάρχουν προβλήματα και σε ό,τι αφορά την δημοκρατική λειτουργία αυτών των χωρών και τη διοργάνωση δημοκρατικών εκλογών. Μέχρι στιγμής, στην περίπτωση Καμπόζη για παράδειγμα, είχαμε την ευκαιρία επανειλημμένης παρατήρησης εκλογών μετά από πρόσκληση της καμποτζενής κυβέρνησης. Οι εκθέσεις ε, ήταν αρκετά επικριτικέ παρόλο που διαπίστωσαν πρόοδο. Άλλε χώρε όμως είτε δεν διοργανώνουν καθόλου εκλογές, είτε οι εκλογές τους δεν είναι δημοκρατικές. Στην Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την παράταση της ισχύω ε, του έκτακτου διατάγματος σε οκτώ επαρχίες και στην Μπαγκόκ, υπάρχει περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Οπότε το τοπίο είναι αρκετά περίπλοκο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο φίλε Πανάμας, που είναι υποδιευθυντής ε, της ομάδας του τμήματος για την Ανατολική Ασία. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για να πω ότι σημεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ, συλλήψεις και καταδίκες οπαδών των οργανώσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως επίσης και όχληση ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων που έλαβαν χώρα στους τελευταίους μήνες και αντιβαίνουν με όλη την πολιτική μεταρρυθμίσεων και ανοιγμάτων των τελευταίων ετών στο Βιετνάμ κατά το διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ στις 25 Ιουνίου στο Ανόη οι βιετναμικές αρχές ε, έκαναν ε, κάποιες χειρονομίες ε, <coughs> κατά τις διαπραγματεύσεις δηλαδή υποδέχθηκαν παρατηρητές από τα Ηνωμένα Έθνη στη χώρα και η επέτειος των 35 ετών από την ανεξαρτησία του Βιετνάμ στις 2 Σεπτεμβρίου μπορεί να οδηγήσει σε μια αμνηστία, απολευθέρωση ορισμένων ε, φυλακισμένων και ελπίζουμε ότι αυτή η αμνηστία θα ισχύσει και για αντιρρήσεις συνείδησης. θα συζητηθεί και με τον κύριο Ζέγκ, τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα έρθει τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητώντας τη νέα συμφωνία συνεργασίας με το Βιετνάμ κατέστησε σαφές στις βιετναμικές αρχές ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία χωρίς να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα εργασίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εν του μελλοντικού συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βιετνάμ το Σεπτέμβριο έχουμε μία συρρήκνωση ε, καθαρά νευρικού χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για κάτι το συστημικό. Ξέρω ότι το Σεπτέμβριο τα μέλη της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής με την ΑΣΕΑΝ θα πάνε στο Βιετνάμ το Σεπτέμβριο και σας ενθαρρύνω να διαμορφώσετε κι εσείς την άποψή σας. Για το Λάος ανησυχούμε ιδιαίτερα για τους ε, περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση, ε, για την ε, κακομεταχείριση της κοινότητας Μποντ. Και οι λαοτιανές αρχές εν ώψη του μελλοντικού διαλόγου του Λάος θα συζητήσουν, θα μας αναφέρουν σχετικά η συνάδελφος η αρμόδια για την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να ανάψετε το μικρόφωνο σας. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σχετικά με την Καμπότζη. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έναν τελεχή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οργανώσαμε και θα οργανώσουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα σεμινάριο για τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε και ένα διάλογο στην Κοινή Επιτροπή. Έχουμε μια υπομάδα εργασίας που θα συνεδριάσει τον Οκτώβριο και θα εξετάσει συνολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευκυβερνησία στην Καμπότζη. Εμείς ε, υποστηρίζουμε, κάποιος αναφέρθηκε εδώ το δικαστήριο των κόκκινων ε, ΚΜΕΡ, ε, η κυρία Ρίτσαρτσον ανέφερε προβληματικές διαφθοράς στα πλαίσια αυτού του δικαστηρίου ανησυχούμε ιδιαίτερα. Εξετάσαμε το θέμα και με τα Ηνωμένα Έθνη και από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η προβληματική βρήκε μια λύση που μας ικανοποιεί πλήρως. Στα πλαίσια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθήσαμε και ετοιμάσαμε με τα κράτη-μέλη την ε, περιοδική ε, έκθεση και θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί. Η αντιπροσωπεία της ΑΣΕΑΝ πήγε τον Μάρτιο στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη και νομίζω ότι η έκθεση θα ακολουθηθεί και από μέτρα τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης που αναγνώρισε ορισμένες δυσκολίες σε ορισμένους τομείς και κυρίως όσον στις προβληματικές που αφορούν στην ελεύθερη έκφραση θα συνεργαστούμε και με την κυβέρνηση αλλά και με την κοινωνία των πολιτών ε, στην Καμπότζη που είναι ιδιαίτερα δυναμική. Έχουμε πάνω από χίλιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, οι οποίες εργάστηκαν μετά από την ε, περίοδο των κόκκινων χμέρ και που βοήθησαν αυτή τη χώρα να πάρει το δρόμο της δημοκρατίας. Για την Ταϊλάνδη σύντομα εμείς ε, λυπηθήκαμε ιδιαίτερα με τα επεισόδια του Απριλίου και του Μαΐου. Η Κατρίνα Άστον ε, έκανε δηλώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρόμαστε για τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για τη συμφιλίωση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την ε, διαδικασία και πρέπει να υπάρξει ένας επικοδομητικός και ενεργητικός διάλογος όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Επίσης ε, σημειώσαμε και τη δέσμευση της θελανδικής κυβέρνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ότι είναι πολύ θετικό γιατί έθεσε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προτεραιότητα θα συμμετέχει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ η Ταϊλάνδη και ελπίζουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος, ε, του σχετικού προγράμματος θα λάβει και τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν στην ελεύθερη έκφραση για τα έκτακτα δια για το διέκτακτο διάταγμα, συγγνώμη. Για τους ε, πρόσφυγες Κμόγκ. εμείς ε, ανησυχούμε επίσης. Και με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης και με την κυβέρνηση του Λάος εξετάσαμε το πώς γίνεται ο επαναπατρισμός αυτών των προσφύγων και ζητήσαμε να επισκεφθούμε τα στρατόπεδα προσφύγων. Για τους ε, βυρμανούς πρόσφυγες ε, συζητάμε με την Ταϊλανδική κυβέρνηση για να έχουμε μια υφόρο ανάπτυξη και όχι απλώς ε, να υποστηρίζουν με μόνο την συντήρηση αυτών των προσφυγικών στρατοπέδων στην Ταϊλάνδη Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς μακροπρόθεσμα μπορούμε να έχουμε μια άλλου είδους εξέλιξη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είδαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ε, αυτές και έχουμε και πολλές χρήσιμες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση, για σχόλια και ερωτήσεις. Κυρία Κιλνίλσεν ζήτησε πρώτο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία πολύ συγκεκριμένη περίπτωση διότι η εκπρόσωπος ε, του, της πρεσβείας του Βιετνάμ αμφισβήτησε τις πληροφορίες που διαθέτουμε εδώ. Έχω μια συγκεκριμένη όμως πληροφορία, την οποία γνωρίζω προσωπικά ως εκλεγμένη της, δυτικής, ε, της περιφέρειας της Δυτικής Γαλλίας και όλοι το ξέρουν δηλαδή και το γράφει και ο τύπος. Πρόκειται για έναν φοιτητή, ο οποίος ε, ήταν πέντε χρόνια ε, στο, στη Γένα, ε, στις εφαρμοσμένες ε, θετικές επιστήμες. Ε, έχετε εδώ και το, τη φωτογραφία του. Λοιπόν, πήρε ένα πολύ καλό πτυχίο, με καλούς βαθμούς, θα έβρισκε και δουλειά στην Γαλλία πολύ εύκολα. Αυτό το, αυτός ο νέος αγαπάει τη χώρα του και θέλησε να γυρίσει στη χώρα του για να βοηθήσει με τις γνώσεις του στη χώρα του. Δυστυχώς όμως είναι ένας ειρηνιστής ε, ε, δημοκρατικός blogger και ίδρυσε και την Ένωση ε, των νέων Βιετναμιτών για την Δημοκρατία. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 7 χρόνια φυλακή τον προηγούμενο Ιανουάριο γιατί θέλησε από ό,τι φαίνεται να ανατρέψει τη λαϊκή κυβέρνηση. Τώρα, στην περιοχή μου που αγαπάει το Βιετνάμ, εγώ ήμουνα αναπληρώτρια δήμαρχος της ΑΓΕΝ και ήμασταν η πρώτη πόλη στη Γαλλία που το 1992 υποδεχθήκαμε ε, μια βιετναμική ε, αντιπροσωπεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ είμαι συνδεδεμένη και με την πόλη της ε, Τουέ. Εμείς αγαπούμε το Βιετνάμ, τους ιατρούς, τους δασκάλους, τους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με, το, με τη ΟΕ και την ε, περιοχή ε, του ΟΕ. Αγαπάμε λοιπόν το Βιετνάμ, δεν είμαστε εχθρικοί ε, έναντι του Βιετνάμ. Υποστηρίζουμε αυτόν τον νεαρό διότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί φυλακίστηκε πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι δυστυχώς μόνο μόνος. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες εδώ, πρόκειται για συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί νέοι Βιετναμέζοι οι οποίοι έκαναν λαμπρές σπουδέ στην Ευρώπη και επιστρέφουν στο Βιετνάμ γιατί θέλουν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της χώρας τους. Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς συγκλονιστήκαμε με τις καταδίκες αυτές στο Βιετνάμ. Και κυρία Κιλίνου, εσείς ξέρετε αυτές τις υποθέσεις από τη Γαλλία. Θα τις σχολιάσει η πρέσβης, ο κύριος Στάνοκ. Εδώ και χρόνια ε, στυλιτεύω την καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ε, δύο βάναυσες ε, κομμουνιστικές χώρες, Βιετνάμ και Λάος. Έχουμε πολλές, πολλούς ε, εξόρους από τις χώρες αυτές και πρότεινα το Τεκουαντού για, για τον Νόμπελ Είναι επιφανή ε, αντιφρονών από το Βιετνάμ. Φυλακή, είναι στη φυλακή εδώ και 30 χρόνια και. Και μάλιστα ε, είδαμε τη βάναυση μεταχείριση των ε, καθώς και τη δίμευση, την αφαίρετη δίμευση των περιουσιακών στοιχείων και της Καθολικής Εκκλησίας και της ε, Ενωμένης Βουδιστικής Εκκλησίας. Για το Λάος ξέρουμε πώς υποφέρουν οι Χμόγκ, ε, που προσπαθούν να αντισταθούν στο, στο κομμουνιστικό καθεστώς. Υπέστησαν βασανιστήρια και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για αυθαίρετες εξοδικαστικές ε, εκτελέσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν την έκκληση προς την κυβέρνηση της Ταϊλάδης να μην εκδώσει τους ε, πρόσφυγες ΚΜΟΝΚ που κατά τη γνώμη μου θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ αβέβαιο πεπρωμένο για να μην πω ε, φρικτό στο Λάος Παλιά το Λάος ήταν ειρηνική μοναρχία και τώρα έχει γίνει μια απομονωμένη και βάναυση κομμουνιστική δικτατορία. Έχει φυλακίσει πολλούς ε, αντιφρονώντες και μάλιστα και πολλούς ηγέτες του φοιτητικού κινήματος του 1999. Για την Καμπότζη δεν ξέρω τόσα πολλά πράγματα. Χαίρομαι για την καθυστερημένη μένα, αλλά τουλάχιστον ε, ε, σύσταση του Μικτού Δικαστηρίου προκειμένου να εκδικάσει περιπτώσεις ε, γενοκτονίας των ε, Ερθρών Χμέρ. Υπήρχε μια δικία τα τελευταία χρόνια και ατιμορρησία που οφείλεται στη διαφθορά της κυβέρνησης αλλά επειδή έχει περάσει πάρα πολλέ χρόνε, είναι δύσκολο να συλλεχθούν τα τα τεκμήρια για να καταδικαστούν, να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι πέτοι. Και στην Καμπότζε εξακολουθούν να, να σειραίουν απειλέ για κακομεταχείριση εκ μέρου αστυνομία, παρόλο που η Καμπότζη έχει υπογράψει πολλέ διεθνεί συμβάσει και του ΙΕ κατά των βασανιστήριων. Η Επιτροπή ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιοχή αυτή και καταδικάζει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Κύριε θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλες και όλους που μας προσέφεραν τόσες πολλές πληροφορίες. Τι να προσθέσει κανείς. Πάντως μου ήρθαν δύο ιδέες ή συστάσεις για την κατάσταση στο Βιετνάμ. Η κυρία Κιλνίλσεν έδωσε κάποια παραδείγματα. Ο ίδιος ο πρέσβης είπε ότι, ή μάλλον, είπε ότι γίνονται προσπάθειες βελτιώσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εθνική επέτειο στο Βιετνάμ στις 2 Σεπτεμβρίου και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας είπε ότι προτίθεται να απολύσει 25-30 ε, κρατουμένους στα πλαίσια γενικής αμνηστίας. Από τις προφορίες που έχω από μη κρατική οργάνωση δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα αυτά πολιτικοί κρατούμενοι. για παράδειγμα άνθρωποι όπως ο νέος τον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κιβ Νίλσεν, αλλά και άλλοι blogger. Και εσύ, κυρία Χάουταλα, και ο πρόεδρος Μπούσεκ θα μπορούσατε ίσως να γράψετε μια επιστολή, γιατί θα μπορούσατε να τους γράψετε πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου, ώστε στους ανθρώπους που χορηγείται αμνηστία να περιληφθούν και αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτή είναι μια σύσταση προς ε, σας ή προς τον πρόεδρο Μπούσεκ. Επίσης τον Σεπτέμβριο έχουμε νομίζω δύο περίοδους συνόδου στο Στρασβούργο. Ίσως μπορούμε να συντάξουμε ένα είδος ε, ψήφισμα για από τις βαρύτερες ε, περιπτώσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων που ακούσαμε εδώ. Ίσως ένα κατεπήγον ψήφισμα για τους ε, ε, για τα πρόσωπα που έχουν επαναπατριστεί στο Λάος από την Καμπότζη. Γιατί η κατάσταση δεν ξέρουμε ακριβώ ποια είναι. Κανείς δεν μπορεί να πάει να επισκεφθεί τα στρατόπεδα αυτά. Οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο πολύ σε απομόνωση και το θέμα βέβαια έχει χαρακτήρα επίγοντα. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τις συστάσεις σας. Ακούσαμε και από τον κύριο Τίμανς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλεί για την δυνατότητα να απολυθούν από τις φυλακές ε, με ευκαιρία της, εθνική, της εθνικής επαιτίου και πολιτική κρατωμένη. Πριν επανέλθουμε στην κυρία Ρίτσαρτσον, θα ακούσουμε την κυρία Γκόμες. Υποστηρίζω τα όσα είπε η κυρία Κιλνίλσεν. Το ενδιαφέρον και η ανησυχία μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές, Καμπότζη, Λαός, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη, ε, απηχεί το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για τους λαούς της περιοχής. Εγώ έχω ταξιδέψει πολύ στην Ινδονησία και είχα εγκατασταθεί κάποιο διάστημα εκεί. Και έχω ε, απεριόριστο θαυμασμό και πραγματική αγάπη για τους ε, ανθρώπους εκεί που εργάζονται σκληρά για, ε, έχω μεγάλο θαυμασμό για την επινοητικότητα των ανθρώπων και για τον πολιτισμό που είναι δικός τους. Και βλέπουμε στην Ερδονησία, για παράδειγμα, πρόοδο με την καθίδρυση της Δημοκρατίας μετά την πτώση του Σουχάρτο το 1980 αλλά δεν βλέπουμε παρόμοια πρόοδο σε άλλες χώρες. Και αυτό έχει σχέση με το είδος καθεστώτων που έχουν εκεί. Και στην Ταϊλάνδη βλέπουμε και οπισθοδρόμηση. και έχοντας υπόψη τις δεσμές που έχουμε αναλάβει και προδεκατιών στην Ευρώπη για να οδηγήσουμε σε τέλος ε, τον πόλεμο του Βιετνάμ, θαυμάζω απεριόριστα τον λαό του Βιετνάμ. Και λυπούμε για την καταπίεση την οποία υφίσταται και που πραγματικά δεν τους αξίζει. Θα συμφωνήσω με τις συστάσεις της κυρίας Λοχμπίλερ. Να γράψετε εσείς, κυρία Πρόεδρε, μια επιστολή. Θυμίζοντας την εθνική επέτειο του Βιετνάμ. Και να συντάξουμε και ιδιαίτερα ψηφίσματα γι' αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Γκόμες με τα λόγια της αυτά απηχεί τα συναισθήματα όλων μας. Όλοι πραγματικά εκτιμούμε και θαυμάζουμε τα επιτεύγματα των λαών αυτών και βέβαια είναι τεχνητός ο τρόπος με τον οποίο συνδέουμε την, ε, τις τέσσερις αυτές χώρες. Γίνεται για λόγους πρακτικούς. Βλέπω ότι η κυρία Δεργά θέλει να λάβει το λόγο και η Δεργιά, συγγνώμη, θέλει να λάβει το λόγο και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε. Μα μου κλέψατε τα λόγια από το στόμα κυρία Πρόεδρε, διότι αυτό το οποίο ήθελα να πω ακούγοντας και τι είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι πραγματικά κάπως τεχνητό το να εξομοιώνουμε όλες αυτές τις χώρες. Η κατάσταση διαφέρει πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν πρέπει να διαμορφωθεί άποψη ότι εμείς ε, ε, τα έχουμε με μία χώρα πιο πολύ από ότι με την άλλη. Οι χώρες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και όπως είπε και η κυρία Γκόμες, έχουμε χώρες που έχουν κάνει σημαντική οπισθοδρόμηση και χώρες που καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και για τη γενική έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέξουμε τις πραγματικές προσπάθειες που γίνονται και να λαμβάνουμε υπόψη την, πραγματική προβληματική της κάθε χώρας αλλά και τη διαφορά της μίας με την άλλη γιατί η κατάσταση διαφέρει πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Ευχαριστώ κυρία βερσέ. Ευχαριστώ. Κυρία Ρίτσαρτσον, πώς βλέπετε τη συζήτηση μέχρι τώρα. Πόσα λεπτά έχω, δύο. Ε, don't speak. Καλά, θα, θα τα πω γρήγορα. Ναι, αλλά μην μιλάτε πολύ γρήγορα. Θα προσπαθήσω. Για το Λάος. Η ιδέα του ψηφίσματος στο Στρασβούργο είναι πολύ καλή και σας ενθαρρύνω να την υλοποιήσετε. Για την Καμπότζη για το δικαστήριο για τους Ερθρούς Χμέρ. Πραγματικά είναι απίστευτο να ε, υποστηρίζει κανείς ότι τα θέματα πολιτικής παρέμβασης ή δωροδοκίας έχουν επιληθεί. Όχι, με αφήνει ευρώτητη μια τέτοια δήλωση ότι έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα. Για την Καμπότζη. Σίγουρα η Καμπότζη διοργάνωσε πολλές εθνικές εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιχαρακώνει και τις δημοκρατικές αξίες και τους δημοκρατικούς κανόνες. Γιατί έχουμε την ίδια κυβέρνηση από το 1994. Από το 1984 και έχουν γίνει και συστηματικές νοθείες των εκλογικών αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά την ε, ύπαρξη των μέσων μαζική ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση βρίσκονται υπό έλεγχο τη κυβέρνηση. Ε, ασκείται κρατικό έλεγχο σε, στα μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχει πολυμορφία δηλαδή ούτε στον τύπο ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Επίση, ε, για το ICCPR και την Οικουμενική Διακήρυξη θα ήθελα να σας εθαρρύνω όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής να ξαναδιαβάσετε τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Παρισιού το 1991 και να θυμηθείτε τι προτάσεις έγιναν στην καμποζιανή κυβέρνηση. Είναι σημαντικό συγκριτικό κανόνα. Άλλη Καμπότζη σήμερα και άλλη Καμπότζη από του Ερυθρού Μέρ ή σε άλλη περίοδο. Και έχουν αναλυφθεί πολλέ υποσχέσει. Για το Βιετνάμ τώρα, Μακάρι να μου στείλει η Βιετναμέζικη κυβέρνηση μια διεξοδική ε, ανάλυση και σχολιασμό των δικών μας εκθέσεων. Επίσης, ότι αφορά την ελευθερία έκφραση στο Βιετνάμ, αν ε, τη σέβεται πραγματικά η κυβέρνηση, τότε γιατί εξέδωσε πέρυσι την ε, ε απόφαση 97 που περί ορίζει τις έρευνες των ε, διεθνών οργανώσεων σε 370 θέματα που έχουν προεγκριθεί από την κυβέρνηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρέσβη. Πιστεύετε ότι η Εξεταστική Επιτροπή που εξεχνιάζει τα εγκλήματα από τον Απρίλιο είναι καλή ιδέα. Εμείς φοβόμαστε ότι αν η Επιτροπή αυτή δεν ε, απαρτίζεται από ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών εκπροσώπων, δεν θα εκδώσει αμερόληπτα και παραδεκτά συμπεράσματα, γιατί είναι χαρακτηριστική η σύνθεσή της και ο τρόπος του και η μεθοδολογία της. Θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση. Σας ευχαριστώ. Φυσικά θα ήταν χρήσιμο να ξαναδώσουμε το λόγο στους πρέσβεις για απαντήσεις, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Γι' αυτό οι, συνεχι... οι συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν μεταξύ σας και μέσω των υπηρεσιών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, ε, ζήτησαν το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση ένα μέλος από την κοινότητα Μπατνακ και κάποιον από το Βιετνάμ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πρώτος στον εκπρόσωπο της κοινότητας Batnam ε, για δύο λεπτά για να μας ε, κάνει μια σύντομη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία αυτή για να μιλήσουμε στην Επιτροπή σας εκπροσωπούμε τα αδέρφια μας ε, των βουδιστών μοναχών στο Βιετνάμ που υφίστανται διώξεις ιδιαίτερα από την θρησκευτική αστυνομία του Βιετνάμ και μάλιστα ε, υπέσαν έξω από το μοναστήρι τους από αστυνομικές δυνάμεις και δεύτερη φορά διαλύθηκε, ε, διαλύθηκε και εκδιώχθηκαν από το ναό που, όπου ένα άσυλο. Τώρα, τους τελευταίους έξι μήνες ε, βρίσκονται ε, εγκαταλελειμμένοι και δεν μπορούν να βρουν πουθενά καταφύγιο. Ζητούμε την υποστήριξη της Επιτροπής. Ε, θέλουμε απλώς να ε, τους επιτρέπει να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία τους, ε, την κατανόηση, τη συμπόνια τους. Είναι η μόνη τους έκκληση. Έχω μαζί μου ε, αυτόπτη μάρτυρα όλων αυτών των γεγονότων που έλαβα χώρα στο Βιετνάμ πριν από λίγες εβδομάδες και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Τάι Χάι από το μοναστήρι της, του Μπατνιάμ για να σας ε, πει δύο λόγια. Σας ευχαριστώ που μας ξαναδίνετε το λόγο. Και την περασμένη φορά που ήρθα ζήτησα τη βοήθειά σας και την προστασία σας για τους αδερφούς και αδερφές ε, στο Βιετνάμ που υπέστησαν ε, επιθέσεις. Γιατί υπήρχαν απειλές για τη ζωή τους. Σήμερα όμως ε, έχω ένα νέα ότι παρά τις διώξεις Κανείς δεν έχασε ούτε την πίστη του, ούτε την ελπίδα του. Παρά τις, α, τις συνεχείς πιέσεις και παρά την άσκηση βίας και ευτυχώς κανένας δεν έχασε τη ζωή του. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ τους ε, συμπολίτες μου, αγαπώ το λαό της και εκτιμώ ιδιαίτερος τις προτάσεις που κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και ξανά για να συζητήσω την υποστήριξή σας, την υποστήριξη για την κυβέρνηση, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση και να προστατεύει τους αδερφούς και αδερφές μας που υφίστανται διώξεις. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια προς την ε, κυβέρνηση. Εκπροσωπώ τους αδερφούς και αδερφές από το μοναστήρι του Μπακνιάμ. Είμαστε νέοι μοναχοί και έχουμε αφιερώσει όλη μας τη ζωή μας στην άσκηση της λατρείας σε ειρήνη και με απόλυτη αποκήρυξη της βίας. Σας έχουμε προσκαλέσει πολλές φορές ε, για συνομιλίες και επικοινωνία, ώστε να καταλάβετε και να υποστηρίξετε τις ελπίδες μας και την πίστη μας και το σκοπό μας. Αλλά δυστυχώς ε, η φωνή μας δεν ακούστηκε, ούτε έγιναν κατανοητά τα αιτήματά μας. Και σήμερα, μπροστά σε αυτή την διεθνή οικογένεια, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να εκφράσω αυτή την επιθυμία μου, την επιθυμία των ε, νεαρών μοναχών, να τι έχουν τις προστασίες και τις κατανόησης από την κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι χωρίς την προστασία και την κατανόηση από εσά, από την κυβέρνησή μας, θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες μας, τις επιθυμίες μας, τους πόθους μας και να ζήσουμε ειρηνικά και με αγάπη και να υπηρετήσουμε το λαό μας με ειρήνη και αγάπη. Ευχαριστώ. Thank you very much, you, indeed. Σας ευχαριστώ πολύ και έχετε την απόλυτη υποστήριξή μας, λέει η πρόεδρος Χάουταλα. Άλλη μια χώρα για δύο λεπτά. Καλώς ορίζουμε τον κύριο Χάρης Αζάρ από μια οργάνωση της Ινδονησίας και τον παρακαλούμε να λάβει τον λόγο για δύο λεπτά. Η οργάνωσή του που έχει το όνομα Κόντρας ε, σημαίνει, σημαίνει την ε, οργάνωση που ε, υποστηρίζει τα θύματα παραβιάσεων ανθρώπων δικαιωμάτων και εξαφανίσεων. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κ. Γκομές προηγουμένως, η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ινδονησία έχει βελτιωθεί. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται επιθέσεις. Ένας ε, ακτιβιστής μας κατά της ε, διαφθοράς έπεσε θέμα ξυλοδαρμού πριν από λίγες μέρες. Στην Πάπουα η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κυρίως ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την υγεία ε, επιδεινώνεται. Επίσης, η ατιμορρησία των δραστών εξακολουθεί ε, να κυριαρχεί, για παράδειγμα για τις ε, παραβιάσεις που έγιναν στο Άτσε. Θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σημαντικά βήματα στην εξωτερική πολιτική και να αναζητήσει τη συνεργασία με την κυβέρνηση της Ινδονησίας που να την οδηγήσει να βελτιώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, η CSO πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία και μέσα στα πλαίσια της ε, διακυβερνητικής επιτροπής της ASEAN. Σας ευχαριστώ. Uh, Κύριε Χάουταλα, σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Μου φαίνεται σωστό να δώσουμε ε, τον λόγο στον κύριο Γκόμες. Ε, στην κυρία Γκόμες, συγγνώμη, ε, που είναι και πρώην πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ινδονησία. Υπάρχουν, πραγματικά ευχαριστώ για το που μου το λόγο, σημαντικές πρόοδοι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα συνεργασία με την διεθνή κοινότητα είναι πολύ σημαντική. Πριν από λίγα χρόνια δηλητηριάστηκε σε μια πτήση προς την Ολλανδία ο Μουνίρ, ο οποίος ήταν και γνωστός μου, και ήταν επικεφαλής του Κόντρας αυτή τη οργάνωσης που προσωπεί εδώ ο κ. Σαζάρ και που όπως είπα δολοφονήθηκε με την ε, άμεση συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών της Ινδονησίας. Η χείρα του θα έρθει να μας δει στο Σασβούργο. Ε, ο Μουνίρη ήταν μια πραγματικά εκπληκτική προσωπικότητα και αποτείω οφόρο τιμή στη μνήμη του και σε όλα τα πρόσωπα που αγωνίζονται στην Ινδονησία υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και η κατάσταση στην Πάπουα είναι τελικά, α, ε, συμφωνώ και εγώ, πάρα πάρα πολύ δύσκολη και η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Η Ινδονησία ασφαλώς είναι μια χώρα που πρέπει να την εξετάσουμε προσεκτικά στην μελλοντική μας εργασία. Δεν είχαμε χρόνο σήμερα να εξετάσουμε τον περιφερειακό μηχανισμό προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΑΣΕΑΝ. Ίσως μπορούμε να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό κάποια άλλη φορά και ένα άλλο θέμα που εφήγει μόνο ε, λίγο είναι η διάσκεψη τον Οκτώβριο του ΑΣΕΜ όπου θα συμμετέχουν, θα συμμετέχουν οι διάφορες αυτές κυβερνήσεις και θα δοθεί ευκαιρία να συνεχιστούν οι διαβουλεύσει και, και επαφές μεταξύ και βουλευτών και ε, προσώπων μη κρατικών οργανώσεων. Ευχαριστώ λοιπόν όλε και όλου για τι σημαντικέ πληροφορίε που δώσατε και ελπίζω τα ανθρώπινα δικαιώματα να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη των χωρών σα και στην εξέλιξη των σχέσεων τη Ένωση μαζί σα. Τώρα, με χαρά μου θα έρθω στο υπαριθμό 6 για την ε, ακρόασή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Μετά από τον τελευταίο γύρο της 29ης έκτου στη Μαδρίτη των ε, συζητήσεων μεταξύ Ένωσης και Κίνας και φαίνεται πως θα γίνει αργότερα και μια διάσκεψη κορυφής Ένωσης Κίνας. Είναι λοιπόν σωστό να συζητήσουμε ξανά το θέμα. Χθε τα μέλη του Διευρυμένου Προεδρείου της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συζήτησαν με αξιωματούχους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα προορίσματα από αυτό το τελευταίο διάλογο, τον τελευταίο γύρο διαλόγου Ένωσης Κίνας και τα μέλη είχαν και πρόσβαση στην μελέτη αξιολόγησης του διαλόγου όπου διαπιστώσαμε ότι χρειαζόμαστε καταβολή εντονότερων προσπαθειών. Υπήρξαν λοιπόν ορισμένες, ορισμένα θετικά σημάδια, κάποιοι μηχανισμοί για την παρακολούθηση των βασανιστερίων και επίσης μια δημόσια συζήτηση για δύσκολα θέματα στην Κίνα που φαίνεται ότι σε πολλούς τομείς δείχνει αυτή η συζήτηση ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων στην Κίνα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε με μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο οι ατομικές περιπτώσεις λοιπόν, είναι οι περιπτώσεις οι οποίες απηχούν μια ε, γενικά ε, ε, εξαιρετικά επιδεινωμένη κατάσταση στην Κίνα. Ο Λιου κρατήθηκε και φυλακίστηκε, είναι ο συντάκτης του Μανιφέστου του 2008, Καλ Σισέγκ, γνωστός ε, συνήγορος και υπερασπιστή ανθρώπινων δικαιωμάτων εξαφανίστηκε και επανεφανίστηκε και ο Χουτζιάρ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή βραβευτή με το βραβείο Ζαχάροφ ενώ κινδυνεύει η υγεία του. Να λοιπόν λίγα μόνο παραδείγματα για το τι συμβαίνει εκεί. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τις ειδήσει που ακούμε για τις συνεχιζόμενες βίες διώξεις σε βάρος των ειρηνικών φιλιρινιστών οπαδών του Φαλουνγκόγκ. Τώρα, έχουμε έναν αριθμό ομιλητών. Θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από τον Λόρδο Ντέβερσον της Βουλής των Λόρδων και που είναι και μέλος της Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βουλής των Λόρδων και θα μιλήσει για την πιο πρόσφατη έκθεση που επιγράφεται Stars and Dragons. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ως πρώην Ευρωβουλευτής, με χαρά μου ξαναβρίσκομαι στο κτίριό σας. Να πω λίγα λόγια για την έκθεσή μας για την Κίνα, που ίσως σας φανούν προφανή, αλλά είναι σημαντικά πάντως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα είναι πολύ σημαντικά, διότι πρόκειται εν τέλει για 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα στην Κίνα και πραγματικά το ένα τέταρτο του συνολικού ανθρώπινου πληθυσμού. Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγής κινέζικων προϊόντων. Οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Κίνας ανάγονται στο 1985 όπου έγινε, συνάφθηκε η πρώτη συμφωνία για εμπορικές σχέσεις και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία συνεργασίας. Από το 2003 άλλαξαν δραματικά οι σχέσεις μετά από την άρση του αποκλεισμού εξοπλισμών μετά το Tiananmen μέν εν τελικά, δεν έγινε μετά από το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι ε, είδε και την Ευρώπη η, η, ε, η Κίνα. Τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Κίνα δεν μπορεί να πει κανεί ότι συνέβαλαν στην πρόοδο του κινέζικου λαού. Και ακόμη και στα 1990 η μεγάλη Βρετανία απεχώρησε από το Χονγκ Κόνγκ όπου δεν είχε και εκεί πάρα πολύ θετική ιστορία. Η Κίνα συμμετέχει βέβαια, είναι ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρεί πάντως ότι η κυριαρχία της είναι σημαντική και οι εσωτερικές της υποθέσεις είναι δική της υπόθεση. Εκεί βρίσκονται και κάποιες δυσκολίες μεταξύ ε, των νοοτροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα. Η έκθεση μας βασίστηκε στο γεγονός ότι εξετάζουμε στην πραγματικότητα ένα μέλλον ε, θα ανήκει στους G2, δηλαδή στην πραγματικότητα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή θα είναι βασικά η σχέση και η Ευρώπη θα παραγωνιστεί. Θα επανέλθω σε αυτό. Εμείς πάντως θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει και ούτε μπορεί να γίνει. τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την Κίνα είναι ότι υπάρχουν ορισμένε αρχέ όπου η κινητική κυβέρνηση δεν πρόκειται να μετακινηθεί σε αυτέ. Η μία Κίνα, για παράδειγμα, όχι σε σχέση μόνο με την Ταϊβάν, αλλά και για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, Θιβέτ, δηλαδή επομένω ένα κόμμα, και πάντα θα υπάρχει ένα κόμμα στην Κίνα, και το κόμμα αυτό θεωρεί εαυτό ότι νομιμοποιείται με την παροχή των ε, συνθήκων για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου, την μείωση της φτώχειας και ότι αυτή είναι η βασική στόχη του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα. Υπάρχουν όμως τεράστια προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, για παράδειγμα με τον μεγαλύτερο αριθμό θανατικών καταδικών, εκτελέσεων θανατικών καταδικών ανά τον κόσμο, ε, ε, δίκες χωρίς καταδίκες χωρίς δίκες, εκπαίδευση δια του σοφρονισμού και ούτω καθεξής. Υπάρχει πολύ περιορισμένη ε, θρησκευτική ελευθερία, μιλήσατε για το Φαλούν Γκόγκ, αλλά επίσης και η παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Συνεχίζονται τα βασανιστήρια, παρόλο που η Κίνα ε, συνυπέγραψε το 1995 την συνθήκη για τις ε, δημόσιες ελευθερίες δεν την επικύρωσε ποτέ. Τέλος πάντων, συζητήσαμε με τους Κινέζους για όλα αυτά τα θέματα και μας κατέστησαν σαφές ότι από τη δική τους σκοπιά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα ποτέ δεν ήταν τόσο καλά και προχωρημένα τα τελευταία 5.000 χρόνια. Και σας δείχνει βέβαια αυτό πώς βλέπουν, με ποια ευρύτητα βλέπουν όλη αυτή την ιστορική εξέλιξη και θεωρούν ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που έχουν βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά και χαίρουν προτεραιότητας. Εμείς βέβαια διαφωνούμε με την τοποθέτηση αυτή, ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η μεγαλύτερη προσέγγιση του στόχου της χιλιετίας οφείλεται στην κινέζικη πολιτική. υπάρχουν και προβλήματα με ε, τις ομάδες Ρώμα, υπάρχουν προβλήματα με, ε, όπως είπαμε, καταδίκες χωρίς δίκες, με ε, παράνομες απελάσεις κλπ. Συνεχίζει το διάλογος της Ένωσης με την Κίνα. Η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεμονωμένες περιπτώσεις σαφώς έχει αποδώσει. Εμείς καταστήσαμε σαφές ότι οι αξίες, οι ευρωπαϊκές αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σημαντικές και διεθνώς και δεν είναι μονάχα ε, εσωτερικό μας θέμα και βρήκαμε και πολλά και σημαντικά έργα ε, αποκατάστασης κράτους δικαίου και στο περιφερειακό επίπεδο στην χώρα αυτή και προγράμματα συνεργασίας τα οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένα. Αυτά δεν τους φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά ενώ τα βρίσκουν πολύ σημαντικά οι επιτόπου Ευρωπαίοι. Το πρόβλημα τώρα του διαλόγου είναι ότι συχνά είναι περισσότερο τελε, τελετουργικός, είναι περιορισμένος. Υπάρχουν περιορισμοί για το ποιο συμμετέχει στο διάλογο και κυρίως από την κινέζικη πλευρά. Και για την ίδια την Ευρώπη είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολιτική ε, διέρη και βασίλευε από πλευρά της Κίνας που εφαρμόζει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα, ε, μάλλον ε, ε, εξαρτάται πάρα πολύ από το ποιο αρχηγό κράτου κυβέρνηση μίλησε πρόσφατα με τον Δαλάη και ούτω καθεξή. Εμεί θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ επιτυχία στις εμπορικέ σχέσεις με ταξί χωρών μελών και κίνα και τη τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έχουμε παραδείγματα τώρα όπως το Ακμαρσίκ, Ευρωπαίου πολίτου, ο οποίος εκτελέστηκε το ε, πέρσι παρόλη την αντίδραση όλων των χωρών μελών. Προς τα που θα κινηθούμε τώρα. Ασφαλώς δεν υπάρχει ε, χώρος ε, να κάνει διδάγματα, να δώσει διδάγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εργαστούμε και να συνεργαστούμε με αλληλεγγύη και θα πρέπει ε, να επιμείνουμε στις ατζέντες μας, κυρίως για τις συναντήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και για θέματα follow-up. Στο Πεκίνο υπάρχει στην αντιπροσωπεία της Ένωσης μονάχα ένας αξιωματούχος ο οποίος είναι αρμόδιος για ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να ενισχυθεί. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας πρέπει ε, να προχωρήσει, πρέπει επίσης όμως να ενισχυθεί εκεί η διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Κίνα, ενώ η ίδια η Κίνα κάνει προσπάθεια για βελτίωση του κράτου δικαίου και στους άλλους τομείς όπου θα ωφεληθεί εν τέλει ε, ε, η Κίνα από βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Κίνα λοιπόν ναι μεν υπήρξε και είναι η πιο επιτυχημένη χώρα ε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, οι μελλοντικέ σχέσει με τι ΗΠΑ θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Ίσως ε, τώρα η δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων να μας επιτρέψει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Αλλά εν τέλει πάντω το ιστορικό ότι του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα δεν μπορεί να είναι δεκτό από εμά του Ευρωπαίου. Ευχαριστώ, Λόρδε Τέβερσον. Δεν με εκπλήσει που η Επιτροπή σας της Βουλής των Λόρδων ε, εκπώνησε τόσο καταπληκτική έκθεση και δεν με εκπλήσει που ήσασταν και εσείς μέλος και συμμετείχατε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης γιατί ξέρετε τα πράγματα αυτά με πολλές λεπτομέρειες. Και όντως υπήρξε σημαντική πρόοδος της ε, Κίνας σε πολλά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Θα δώσω τώρα το λόγο με ιδιαίτερη χαρά στον κύριο Γουάν Γιανχάη για ένα δεκάλεπτο για πολλά χρόνια έκανε εξτρατεία υπέρ τη υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και μάλιστα ίδρυσε και μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Beijing ICC Inc., ε, Ινστιτούτο Υγείας, αρχική ονομασία τη CIZING. Κύριε Βάνια Χάι, εργαστήκατε επίσης ε, πολλά χρόνια για την ε, καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης για την πρόθεση των δικαιωμάτων των ε, θυμάτων ή των ασθενών του AIDS ή άλλων σεξουαλικά μεταδοτικών ασθενειών, ε, υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων μειονοτήτων. Ε, Προσπαθήσατε να δημιουργήσετε μια αφύπνιση και για τα κοινωνικά δικαιώματα στην Κίνα και μάλιστα το πιο τολμηρό και θαραλέο τμήμα του έργου σας είναι να προωθήσετε δικαιώματα ομοφιλοφίλων στην ε, ε, Κίνα καθώς και των ε, πορνών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το λόγο, για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο έργο μας στην Κίνα, ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμεινο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί συστηματικά την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της ε, πολιτικής ελευθερίας στην Κίνα κατά την ε, σύναψη διμερών σχέσεων με τη χώρα αυτή. Έχω, ε, ανήκω στον τομέα της υγείας και ασχολούμαι με τα θέματα υγείας πάνω από 20 χρόνια, αλλά το Μάιο χρειάστηκε να εγκαταλείψω και πάλι τη χώρα μου και ελπίζω να με βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικώς δικαιούμαι ακόμη να επιστρέψω στην Κίνα, αλλά το πολιτικό κλίμα δεν είναι πρόσφορο για μένα. Για να επιστρέψω στην πατρίδα μου, δεν θα μπορέσω να διαχειριστώ και να ασχοληθώ με τη λειτουργία της οργάνωσής μου. Και μάλιστα διατρέχω τον κίνδυνο και διώξω να από την κυβέρνηση. Το τελευταίο εξάμεινο η οργάνωσή μας βρέθηκε στο στόχαστρο κάποιων κυβερνητικών υπηρεσιών. Εμείς ιδρύσαμε την οργάνωσή μας το 1994, αρχικά ασχολήθηκε με κοινωνικά προγράμματα και το 2002, το Δεκέμβριο του 2002, ο συνάδελφος Χουτζάη, εγώ και κάποιοι άλλοι, ιδρύσαμε και επίσημα και καταχωρήσαμε την οργάνωσή μας ως επιχείρηση, ως εταιρεία. Βέβαια η κυβέρνηση μας υποχρέωσε να αλλάξουμε το όνομά μας, αλλά εμείς ε, εξακολουθούμε να την αποκαλούμε το Ινστιτούτο Υγείας του Beijing. Πολλές οργανώσεις σαν τη δική μας είναι υποχρεωμένες ε, να καταγράφονται ως εταιρείες από άψη φορολογική και εξαιτία των περιορισμών που υπάρχουν για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Κίνα. Το Ινστιτούτο μας ασχολείται με την πρόληψη του AIDS, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν άνθρωποι πιο περιθωριοποιημένοι. Ασχολούμαστε με φιλομεταβατικούς πόρνες, ομοφιλόφιλους, μειονότητες και ασθενείς ε, με AIDS και άλλες μεταδοτικές σεξουαλικά ασθένειες. Μάλιστα, ε, συμμετέχουμε σε ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων που ασχολούνται με το AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώ. Έχουμε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο κίνημα των ομοφιλοφίλων και μάλιστα συμβάλαμε στην αποκάλυψη ενός ε, σκανδάλου με το αίμα στην Κίνα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που πάσχουν από AIDS και ιδιαίτερα τις μειονότητες ε, που βρίσκονται σε πιο ευπαθή κατάσταση των αρκομανών και των ε, ασθενών με AIDS. Το τελευταίο εξάμεινο η οργάνωσή μας υπέστη σοβαρές παρενοχλήσεις από την κυβέρνηση. Και μάλιστα ε, προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε τον εορτασμό της 16ης επαιτίου μας, αλλά για δύο εβδομάδες είχα παρκαρισμένο αστυνομικό περιπολικό μπροστά στο σπίτι μου και μάλιστα σε ένα εργαστήριο ε, που είχα οργανώσει για την προστασία της υγείας των ε, πορνών ε, δεν μπόρεσα τελικά να το διοργανώσω, απαγορεύτηκε και μάλιστα απαγορεύτηκαν ε, Απαγορεύτηκε και στα μέσα μαζική ενημέρωση να παραπέμπουν στο έργο μα ή σε εκθέσει μα. Και μάλιστα κάποιος από το εμπορικό επιμελητήριο του Πεκίνου ήρθε στο γραφείο για να κάνει μια ε, εξέταση των λογαριασμών και μας είπε ότι το όνομα που χρησιμοποιούμε στις ε, δραστηριότητές μας δεν είναι αυτό με το οποίο έχουμε γραφεί επισήμως. Επίσης, το Μάρτιο του 2005, το εκπρόσωπος εφορίας ε, ξεκίνησε μια φορολογική έρευνα στην εταιρεία μας. Ήταν η δεύτερη έρευνα που υπέστημε την τελευταία διετία. Επίσης, η εφορία μας ζήτησε σχεδόν όλα τα έγγραφα εργασίας των τελευταίων 8 ετών. Για παράδειγμα, ζήτησαν όλους μας τους λογαριασμούς, όλους τους οικονομικούς φακέλους και στοιχεία για όλους μας τους συνεργάτες. Κάτι που παραβιάζει την ιδιωτική σφαίρα αυτών των ανθρώπων. στις 30 Μαρτίου έδινα μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Γουαντζό που διακόπη από αστυνομική παρουσία. Και την επόμενη μέρα όλα τα πανεπιστήμια της Γουαντζό έλαβαν εγκύκλιο ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στον αντιφρονούντα Γουανχάι να δίνει διαλέξεις. Επίσης, κάποιος αρμόδιος από την περιοριστική έκανε έρευνα στα γραφεία μας και την περασμένη εβδομάδα Μία εταιρεία που μας βοήθησε να εκδώσουμε εκπαιδευτικό υλικό δέχτηκε έλεγχο από την ε, αστυνομία της περιφέρειας. Βλέπετε ότι γίνονται πολύ συχνά έλεγχοι των δυνάμεων ασφαλεία ε, στα γραφεία μας. Δεν είμαστε η μόνιμη κυβερνητική οργάνωση που με ε, επιθέσεις και πέρυσι η εφορία του Πεκίνου ανέλαβε μια τέτοια πρωτοβουλία κατά πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και μάλιστα πέρυσι συνέλαβε και για τέσσερις μήνες και φυλάκισε έναν επικεφαλής άλλης μη κυβερνητική οργάνωση. Το ίδιο έγινε και με την Oxfam, που δέχτηκε επιθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας. πολλές εταιρείες έχουν απειλέ ε, για μη συνεργασία μαζί μας. Και έγιναν παρεβάσεις και στο δίκτυό μας. Η κυβέρνηση πρόσφατα έχει θετήσει μια νέα πολιτική και προσπαθεί να εμποδίσει τους διεθνείς δωρητές να χρηματοδοτήσουν ε, τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. είναι σαν το firewall που υπάρχει στο ίντερνετ. Ουσιαστικά προσπαθεί να απομονώσει τις τοπικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις από την πρόσβαση σε διεθνή χρηματοδότηση. Και αυτό έχει επηρεάσει τις λειτουργίες ε, και τις δραστηριότητες πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Κίνα. Η Κινέζικη κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, επιτέθηκε και σε άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε θρησκευτικέ οργανώσεις, σε δικηγόρους ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αντιφρονούντες, σε ακτιβιστές εθνικών μειονοτήτων. Προσπάθησε να ελέγξει και το διαδικτύο και εμπόδισε πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις να εκδίδουν ανακοινώσεις μέσω του ίντερνετ. Σε ό,τι αφορά το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα, Κατά τη γνώμη μου, στην, στην πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να βοηθήσει την Κίνα να μεταβεί σε μια κοινωνία σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ήπιο τρόπο. Εγώ ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις επαφές με την Κινέζικη κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική και στρατηγική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στην Κίνα. Θα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει κάποιες στρατηγικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών στην Κίνα και να βοηθήσει την ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα και επίση να έχει διάλογο μαζί τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, έχω καταθέσει και γραπτό κάποιε συστάσει για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δημοσιεύει πληροφορίε και να ζητά σχόλια και πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και επίση να αναμίξει την κοινωνία των πολιτών σε στρογγυλέ τράπεζε ή σε σεμινάρια και διασκέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή μπορεί στα σεμινάρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Κίνας. Εμείς έχουμε ζητήσει συμμετοχή της κυβέρνησης σε τέτοιους διαλόγους. Αλλά η μπορει στα σεμιναρια τη ευρωπαικη επιτροπη να καλει Επιτροπή εμεις εχουμε ζητησει συμμετοχη τη κυβερνηση σε τετοιου διαλογου αλλα η ευρωπαικη επιτροπη μπορει μεσω και των πρεσβειών των κρατών μελών να έχει πολύ πιο εκτεταμένες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στην Κίνα και οι διεθνεί ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που συμμετέχουν στο διάλογο θα μπορούσαν να συνεργαστούν με του ομολόγου του ε, στην Κίνα για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για θέματα χρηματοδότηση, θα πρότεινα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειριστεί ξεχωριστά τη σχέση της με την κυβέρνηση και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη απέτηση για υποστήριξη από ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Θα πρότεινα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το κονδύλιό της για την αρρωγή προς ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω πολλά σχόλια, θα σας δώσω τη γραπτή μου δήλωση. Πάντως η τελευταία μου πρόταση θα ήταν είναι ότι υπάρχει μια πολιτική, ε, η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Χωρίς μια τέτοια πολιτική ε, αντιπαράθεση και ένα πολιτικό ανταγωνισμό, η κυβέρνηση δεν ε, θα μπορέσει να λάβει υπόψη και τη φωνή των πολιτών. Πολιτικά δεν υπάρχει αρκετή πολυμορφία στην Κίνα. Γι' αυτό και θα ήθελα να θαρρύνω την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Κίνα προκειμένου να, να αναπτύξει μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και μια μεγαλύτερη πολυμορφία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε σημειώσαμε τις δυσκολίες και τις παρενοχλήσεις που αντιμετωπίζετε στο σημαντικό έργο σας. Ακούσαμε και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τον διάλογο μεταξύ Ένωσης και Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από εσάς και από τον κύριο, από τον Λόρδο Τέβερσον. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή, αλλά τώρα θα παρακαλέσω την καθηγήτρια Μαρή Χόλτσμαν να λάβει το λόγο, συνολόγο, πρόεδρο της Ένωσης Αλληλεγγύης, του συνδέσμου μάλλον αλληλεγγύης με την Κίνα, η κυρία Χόλτσμαν. Σας ευγνωμονώ που με καλέσατε να μιλήσω σήμερα και είναι μεγάλη μου τιμή που μιλάω με το, μετά τον κύριο Ουάνου Γιανχάη του οποίου την εργασία, τις εργασίες παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια ως παρατηρήτρια και θαυμάζω την αποφασιστικότητά του και το κουράγιο του. Εγώ υποστηρίζω όλα αυτά τα οποία είπε και τις παρατηρήσεις του για την προστακτική ανάγκη που υπάρχει να βοηθήσουμε την, ε, τους πολίτες ε, της ε, Κίνας και βέβαια αυτό το βλέπει με πάρα πολύ ε, κακό μάτι η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Τα τελευταία δέκα χρόνια η κινέζικη οικονομία έχει πετύχει ε, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως ε, που διαφεύγει είναι ότι τα, αυτές οι τελευταίες οικονομικοί πρόοδοι των 30 ετών δεν συναδεύονται από πολιτικές πρόοδους ε, Θυμάστε καλά την Τιαναμέν, ε, τις ε, συλλήψεις ε, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τις καταδίκες σε θάνατο χιλιάδων Κινέζων πολιτών. Πολλοί έχουν καταδικαστεί με, αυθε, με, με αυθαίρετο τρόπο, με, μετά από βασανιστήρια ή ειρηνικές ε, διαμαρτυρήσεις στο Θιβέτ και στο Σίντζαν δεν ε, αποδεικνύουν να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2010, στο ο κύριος ε, Λίλι Μεν, ο οποίος είναι καθηγητής στο Κινέζικο Ιστιτούτο ε, για την κινέζικη ανάπτυξη και τις εξωτερικές σχέσεις και το εξέφρασε αυτά με αυτό με έναν κινέζικο ρόλο που σημαίνει επιφανειακή ελευθερία προς τα έξω αλλά φοβερή, ε, φο, φοβερή αυστηρότητα στο εσωτερικό. Και ο κύριος ε, Λίλι Μέιν λέει ότι κυρίως ε, στο στρατιωτικό τομέα υπάρχει μια γενική συσκότηση των ε, γνώσεών μας για την Κίνα. Λοιπόν, η Κίνα είναι κοινική. Ε, προ, θεωρεί ότι η καταστολή είναι ένα μέσο ελέγχου του πληθυσμού και η χρήση της ε, βίας αυξάνεται συνέχεια διαπιστώνουμε παρεμβάσεις μαφιόζικου χαρακτήρα σε όλες τις κλίμακες της ε, κινέζικης κοινωνίας και αυτές οι παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα βίες. Είναι σαφές ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του ΟΗΕ είχαν κάποιες επιτυχίες στα τέλη του 1990 διότι τότε η Κίνα ήθελε να μπει στην ΠΟΕ αλλά μετά από το 2001 που έγινε μέλος της ΠΟΕ και μετά από το 2008 των Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή στο Πεκίνο οι πιέσεις από τη Δύση σημαίνουν χωρίς κανένα, καμία απάντηση. Ο κύριος Σαμπό έχει καταδικαστεί σε 11 χρόνια φυλάκιση το προηγούμενο φθινόπωρο. Αυτό είναι κάτι το... είναι ένα μήνυμα σαφέστατο και αυτό ήταν και το χριστουγεννιάτικο δώρο που μας έκαναν οι Κινέζοι λέγοντας ορίστε ουσιαστικά τι θεωρούμε εμείς για τις προσπάθειες που κάνετε για να προστατεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα της ε, Κίνας. Ε, στην Κίνα είναι πάρα πολύ προσκολλημένοι ε, όλοι στο, στο ημερολόγιο οπότε αυτή η πράξη καταδίκης ε, δεν έγινε τυχαία εκείνη την ημερομηνία και κάτι ήθελε να πει. Από την άλλη η δυτική κοινή γνώμη έχει τυφλωθεί από την, ε, και τυφλώνεται όλο ένα και περισσότερο από την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και την πρόοδό της και παρά την καλή δουλειά ορισμένων δημοσιογράφων, ευρωπαίων δημοσιογράφων στην Κίνα ε, όλη αυτή η προβληματική κάπου χάνεται ορισμένοι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες τους μίλησαν για προσωπικότητες που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Κίνα το ίδιο και, ορισμέ... και πολλές εφημερίδες έχουν αρχίσει και κλείνουν οι Far Eastern Economic Review για παράδειγμα που είχε έδρα το Hong Kong ε, αναγκάστηκε να κλείσει. Και έχουμε πολλές, ε, πολλά παραδείγματα αυτού του τύπου. Ας πούμε μία ε, μικρή εταιρεία παραγωγής ντοκιματέρ στο Πεκίνο ή παραγωγή, οι παραγωγές χικάρι αναγκάζονται να φύγουν από το Πεκίνο. Λόγω της 20ης επαιτίου της μέν ε, το 2009 η εταιρεία Χικάρη έτυχε τριών ε, ελέγχων όπου κατασχέθηκαν DVD ε, και υλικό των διαφόρων ντοκιμαντέρ και μάλιστα αυτά τα ντοκιμαντέρ πρόκειτο να, να, να, να, να προβληθούν στη Γαλλία και κατάφεραν οι κινέζικες αρχές να παγορεύσουν και την προβολή τους στη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν απόλυτη, σχεδόν απόλυτη λογοκρισία για τα καυτά θέματα, τι έναν μεν και τα λοιπά, αλλά βλέπουμε την Κίνα να παρεμβαίνει με διάφορους ε, λεπτούς ε, τρόπους και στην ε, Δύση για να επιβάλλει λογοκρισία. Έχουμε πολλαπλασιασμό των ε, Κινέζικων Μορφωτικών Ινστιτούτων Κομφούκιους ε, ε, που παίζουν αυτόν τον ρόλο στην Ευρώπη αλλά και, στην, και στα πανεπιστήμια. ορισμένοι συνάδελφοί μου δεν πάνε πια στην Κίνα διότι τους, ε, δεν τους δίνουν θεώρηση και μπαίνουν σε μαύρες λίστες. Εδώ και 15 χρόνια που είμαι και εγώ στη μαύρη λίστα έχω την ελευθερία του λόγου ανεπιφύλακτα αλλά δεν πάω στην Κίνα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για, το, για αυτό το γεγονός αλλά για έναν ε, συνολόγο ε, έχει μεγάλες επιπτώσεις στο επάγγελμά του. Επίσης διαπιστώνουμε σε όλες τις ιστοσελίδες ε, του, στο ίντερνετ να έχουμε επαγγελματίες αντιρρησίες. Ο καθένας μπορεί <clears throat> να φτιάχνει ένα μπλοκ μεγάλο ή μικρό ε, για την Κίνα, για τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες κτλ. Αλλά οτιδήποτε και να γράφετε δίνεται αμέσως απάντηση για να βάλει τα πράγματα για να βάλουν το συντάκτη του blog στη θέση του. Για παράδειγμα γράφετε εσείς ένα blog ότι το τάδε δημόσιο έργο έχει διακοπεί, ε, τότε ε, υπάρχει, θα πιστώσετε ότι αμέσως υπάρχει απάντηση που δικαιολογεί την κατάσταση και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Λέγονται One Mao αυτοί στην ε, Κίνα, δηλαδή είναι οι έμιστοι για να παρεμβαίνουν ε, στα διάφορα μπλόκα. Παίρνουν μισό ευρώ την ώρα. Γουμάου λέγονται λοιπόν. Αυτή η λογοκρισία ταυτόχρονα συνδέεται με τη δυσανάλογη αύξηση πληροφοριών που έχουμε από την Κίνα. Το 2000 το 2009 η Κίνα οργάνωνε την διάσκεψη κορυφή των μίντια και από τότε ξεκίνησαν δισεκατομμύρια για την πληροφόρηση μεταξύ των οποίων και η αγγλόφωνη τηλεόραση, η Συνσημέη η οποία <coughs> ενημερώνει στα αγγλικά εκατομμύρια ανθρώπους. Το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων έχει εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Έχουμε πολύ μεγάλα παραδείγματα. Αυτή η αγγλόφωνη λοιπόν τηλεόραση ε, θα συμπληρώσει τις δρατηριότητες του Κινέζικου Πρακτορείου Σίγουα και ο Κινέζικος πρόεδρος λέει, ο Κινέζος πρόεδρος συγγνώμη, λέει ότι θέλουμε να έχουμε μια παγκόσμια ορατότητα. Κανένας δεν έχει αντιρρήσεις ε, τα, κινέζικα, μέσα ε, μασικής ενημέρωσης να ενημερώνουν την δυτική κοινή γνώμη. Αλλά εκείνο το οποίο βρίσκω απαράδεκτο είναι ότι όποιος άλλος θέλει να πει κάτι του, τον φημώνουν. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να έχουμε περισσότερες εκπομπές στα κινέζικα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτή την προσπάθεια αποπληροφόρησης εκ μέρους των κινέζικων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ καθηγητά Χόλτσμαν. Πραγματικά συναρπαστική η λεπτομερής ανάλυση που μας προσφέρατε και τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα για α, λογοκρισία και οι συστάσεις που κάνατε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος έχουμε τον κύριο Βανσάν Μέτεν που εκπροσωπεί την ε, διεθνή εκστρατεία υπέρ του Θιβέτ και ας μην δυσμονούμε ότι μετά την εξέγερση της 8 Μαρτίου του 2008 εξακολουθούν εκατοντάδες Θιβετιανών να είναι φυλακισμένοι και τα όσα ακούμε για την απίστευτα σκληρή μεταχείριση που τους ε, επιφυλάσσουν και ιδίως όσοι ε, έχουν κάποιο θρησκευτικό αξίωμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Όλοι, όλες οι συζητήσεις που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο για τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Για την κινέζικη υπόθεση, 27 χώρες αντιμετωπίζουν διαφορετικά την Κίνα. Ανάλογα δηλαδή με το τι έχουμε να κάνουμε με την Κίνα, το Θιβέτ ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι θέλει η Ευρώπη, ποιο είναι το στρατηγικό της όραμα, ποια είναι η πολιτική της οραμα ποια ειναι η πολιτικη της στόχοι, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που δεν μπορεί να δεχθεί και να ξεπεράσει. Έχει ορίσει έναν, πρέπει να ορίσει έναν αντιπρόσωπο, ειδικό αντιπρόσωπο για το Θιβέτ, πρέπει να δοθεί ένα καθεστώς στον Δαλάη Λάμα θα πρέπει να γίνει ε, συνάντηση ε, του είπα του εκπροσώπου με τον Δαλάη Η κυρία Άστον όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσει. Αυτό το νέο μέσο θα πρέπει να διαπαιτεί από πολιτικούς και συνεκτικούς ε, στόχους και δεν θα πρέπει να είναι διστακτικός. Η τελευταία μελέτη του Φρανσουά Γκοτμάνα για την ε, κινέζικη πολιτική ε, κάνει μία εύστοχη ανάλυση για την σχέση ΕΕ Κίνας και κάνει προτάσεις λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει συνεκτικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, συντονισμός μεταξύ εθνικών κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάλογος με την Κίνα έγινε το Ιούνιο ε, στρατιωτική συνεργασία, ο ένας διάλογος και ο δεύτερος για τον ελαφρό οπλισμό. Αυτό όμως δεν αντιβαίνει το εμπάργο για τα όπλα που ισχύει. Ε, Δεύτερο, σχέσεις, ε, μακροοικονομικές και εμπορικές σχέσεις και εξωτερικές σχέσεις και εύνομη διακυβέρνηση από την άλλη. Εμείς δεν πρέπει να αποκλείουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις στους άλλους τομείς. Πρέπει να ε, ορίσουμε ε, την απαγόρευση ε, εισαγωγής προϊόντων που κατασκευάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης θα πρέπει πάντοτε εμεί δε να κάνουμε μία αποτίμηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα για τις εμπορικές σχέσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε υπηρεσίες εξωτερικές δράσεις που θα ε, προβληματίζονται για το ρόλο των Ευρωπαίων διπλωματών, για τις μη κυβερνητικές κυβερνήσεις να τους προδώσουμε νομιμότητα. Επίσης ε, θα πρέπει να ε, μιλήσει ο ύπατος, ύπατη εκπρόσωπος για τις πιέσεις που δέχονται τα κράτη-μέλη σχετικά με το Θιβέτ. Στην Μαδρίτη έγινε μία διάσκεψη και δόθηκαν και, και ένας Κινέζος διπλωμάτης εκεί δέλησε να διακόψει την έκθεσή μου. Και εγώ όμως μίλησα για την προστασία των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών διπλωμάτων. Μιλήσαμε επίσης και για την ε, συνεχή καταπίεση των καλλιτεχνών και των ε, διανοουμένων Κινέζων και Θιβετιανών, ε, και η καταστολή επίσης ε, των ε, εκφράσεων εθνικής ταυτότητας των πολιτών του Θιβέτ. Εμείς θελήσαμε να περάσουμε το μήνυμα και να αντιπαρατεθούμε, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος πρέπει ακόμη να φανεί. Έχουμε επίσης και το Human Rights in China, το εμπόδιο για τη λειτουργία ε, αυτής της οργάνωσης είναι οι Κινέζοι, οι ίδιοι οι οποίοι εμποδίζουν τις, ε, τα λόγια να γίνουν πράξη. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να ελέγχει τα πάντα. Οι προσπάθειες λοιπόν είναι καθαρά ε, επιφανειακές. Εμείς δεν γίνονται για παράδειγμα δεχτές οι αιτήσει αμνηστίας για τις θανατικές ποινές. Εμείς επίσης για τις αξιολογήσεις ε, θέλουμε να πούμε ότι η τελευταία ευρωπαϊκή αξιολόγηση δεν δημοσιεύτηκε. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Πρέπει επίσης ε, να έχουμε πάντοτε ε, το προσωπικό αρχείο του κάθε κρατουμεκνού και να συμπληρώνουμε με την κάρτα ε, αυτού του κρατουμένου έναν κατάλογο για να μπορούμε μετά να απαιτούμε την απολευθέρωσή του, να ενισχύσουμε το ρόλο και τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανίσεων, των ομπερογνωμόνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βοηθήσουμε τους, ε, προσπιστές, τους Κινέζους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, να επιτρέπουμε την κυκλοφορία της πληροφορίας μεταξύ των όσων συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις Κινέζων και Ευρωπαίων. Αυτό δεν συνέβη στη Μαδρίτη. Τελευταία σύσταση. Πρέπει να συντονίσουμε την ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών που έχουν διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρία Πρόεδρε, λόγω της ε, αλαζονίας ε, των κινέζικων αρχών απέναντι στις κριτικές της Ευρώπης, <coughs> συμφωνώ με τον Wang Yanhai, ώστε η Ευρώπη να υποστηρίξει τους διανοούμενους της Κίνας και το, το, Θιβέτ, να υποστηρίξει όλες τις νέες αναδεόμενες πολιτικές δυνάμεις για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η σχετική έκθεση που έγινε για το Θιβέτ ΒΕΤ ζητάει να τεθεί το θέμα στην επόμενη αντιπροσωπεία που θα πάει στο ΘΙΒΕΤ. Επίσης, στον προϋπολογισμό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναφέρει και τα σχέδια συνεργασίας και υποστήριξης των εξορίστων Θιβετιανών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέτεν. Μας κάνατε ορισμένες σημαντικές συστάσεις για τον διάλογο και οι τρεις ομιλητές περιλαμβανομένη της καθηγητρίας Χόλτσμαν, με τον δικό της τρόπο, τονίσατε την ανάγκη διαφάνειας στον διάλογο. Μιας και έχουμε την αγαπητή δόκτωρα Ρίτσαλσον της Human Rights Watch κοντά μας, που είναι και η Advocacy Director για την Ασία, θα ήθελα να της δώσω την ευκαιρία να συμμετάσχει πάλι στη συζήτηση Μπορέσαμε πριν βέβαια να ανταλλάξουμε απόψει για τον ε, διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Κίνα σε άλλη ευκαιρία. Έχετε τώρα λοιπόν το λόγο κυρία μου. Οι προηγούμενοι αγορητές κάλυψαν πολύ καλά το θέμα ήδη της ε, κατάστασης ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Θα έρθω λοιπόν εγώ μόνο ε, στους μηχανισμούς των σχέσεων μεταξύ Ένωσης και Κίνας. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί περισσότερο την αξία την οποία αποδίδει η κινέζικη κυβέρνηση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου που είναι και βασική στόχη της Ένωσης. Η πρόκληση για την Ένωση είναι να παρέμβει δυναμικά σε όλες τις ε, ε, σχέσεις της με την ε, κινέζικη κυβέρνηση, κυρίως σε τομείς που είναι σημαντικοί για την κινέζικη κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα ο διάλογος για το εμβόριο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελέσουν ξεκάθαρο και αναπόσπαστο μέρος του διαλόγου μεταξύ Ένωσης και Κίνας. και να υπάρξουν συνέπειες εάν δεν ε, βελτιωθεί η κατάσταση. Στον πιο πρόσφατο γύρο του διαλόγου αυτού διαπιστώνονται ότι, δεν υπάρχουν benchmarks για, τον διάλογο για, τη, για, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπως είπε και ο Λόρδος Τέβερσον είναι αδιαφανής η ε, οι της κινέζικης κυβέρνησης ε, εν προκειμένου και οι πληροφορίες που καταθέτει η ε, κινέζικη κυβέρνηση σε απάντηση ερωτήσεων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος είναι προβληματικός επίσης κατά την έννοια ότι όχι μόνο η δομή του δίνει την ευκαιρία στην κινέζικη κυβέρνηση να συγκρίνει ε, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα με ε, δίθεν παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ένωση, αλλά δίνει και την ευκαιρία και σε άλλα επίπεδα του διαλόγου Ε, μάλλον εμποδίζει άλλους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο διάλογο αυτό και που είναι εκτός κυβερνήσεως να συμμετάσχουν. Σχετικά με το σεμινάριο στην Μαδρίτη, ο σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να συμπληρώσουν τον ε, επίσημο διάλογο. Η τελευταία συνεδρία ήταν καλύτερη, λίγο καλύτερη από προηγούμενες, πρόσφερε στις μη κρατικές οργανώσεις κάπως μεγαλύτερο ρόλο στις συζητήσεις ε, και έγιναν ανταλλαγές απόψεων που δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικές συζητήσεις, αλλά τουλάχιστον κάποιοι μίλησαν μεταξύ τους. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στην κατάσταση, ούτε είναι επαρκής η πρόοδος αυτή που σημειώνω. Εξακολουθούν οι διάλογοι αυτοί να είναι πολύ περιορισμένοι και αυτοί που γίνονται στην Ευρώπη. Η συζήτηση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα προβληματική. Η κινέζικη πλευρά είτε δεν ενδιαφέρεται για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, είτε δεν έχει τη δυνατότητα να δράσει με βάση τέτοιες ε, βέλτιστες πρακτικές. Και είναι και αδύνατο να τους αναγκάσει κανείς να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Εγώ έθεσα μια ξεκάθαρη υποθετική ερώτηση στην Μαδρίτη, πώς θα έπρεπε δηλαδή να λειτουργήσει η διαδικασία και ούτε καν σε αυτό δεν μου απάντησαν. Επίσης πολύ λίγες μη κρατικέ οργανώσεις κινέζικες προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Κάποια από τα βήματα που θα θέλαμε να δούμε για να διορθωθεί η κατάσταση να μην αποκλείεται ή οσδήποτε από το πουλ των Ευρωπαίων ε, εμπειρογνωμόνων λόγω κάποιων ευαισθησιών ευρωπαϊκών ή κινέζικων για το έργο τους. Χρειάζονται Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες που έχουν γνώση για την κατάσταση στην Κίνα και τις πραγματικότητες που σημειώνονται εκεί, να επιτρέπεται στους διεθνείς ε, μη κρατικούς οργανισμούς να συμμετέχουν, benchmarks για τον διάλογο, για να υπάρξουν βελτιώσεις. Για παράδειγμα, ζητήστε να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για την κύρωση της ICCP. Μπορείτε να ζητήσετε για παράδειγμα την απόλυση αντιφρονούντων. Πράγματα τα οποία ζητούν εδώ και, ε, ζητούμε εμείς εδώ και μία δεκαετία. Επίσης, η μετάβαση τώρα στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Εμείς ζητούμε να παραμείνει εστιασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση στις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όποιο και να είναι το αρχικό σας παιχνίδι εντό εισαγωγικών απέναντι στους Κινέζους, οι Κινέζοι θα κάνουν την βέλτιστη προσφορά τους. Και πρέπει να εξετάσετε τις ε, αρχές που διακυβεύονται εφόσον ε, τροποποιηθεί η δομή. Γενικά θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός ο διάλογος ε, να διαρθρώνει, να αρθρώνει δηλαδή τους όρους ε, τους οποίους επιθυμεί να δει να πληρούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση του αποκλεισμού, του εμπάργου δηλαδή του εξοπλισμού. Οι συζητήσει αυτές γίνονται δύο φορέ το χρόνο. Συμφωνώ με τον Λόρδο Τέβερσον και την σύστασή του ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίε για συνεργασία με μια στρατηγική που μπορεί να είναι η επιλογή ορισμένων κοινών στόχων που να ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές ε, και μηχανισμούς επιβολής. Εμείς πολύ ευχαρίστως να σας δώσουμε κάποιες συστάσεις σχετικά με, τα, με το ποια θέματα θα μπορούσατε να επιλέξετε. Και τέλος, η Human Rights Watch θεωρεί ότι η κινέζικη κυβέρνηση όχι μόνο αντιδράσει σε διεθνή πίεση, αλλά ακόμα περισσότερο όταν είναι ε, συντονισμένη η διεθνής αυτή πίεση από πολλές χώρες. Αυτά μπορούν να γίνουν και με πιο δημόσιο τρόπο, με συμμετοχή στις συνεδρίες και ε, εκπροσώπων ε, γνωστών διεθνών οργανώσεων προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων εμπειρογνωμόνων και να προσπαθήσετε να εξέβρετε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να μιλήσετε με μια φωνή για την εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά εξαιρετικές οι συστάσεις σας για την ε, πρόθεση του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σημειώνω επίσης ότι η αδιαφάνεια είναι όντως πρόβλημα και το ότι αποσπάστηκε το νομικό σεμινάριο από το πεδίο του διαλόγου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόκας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα γίνει συζήτηση. Ο κύριος Ρόκας. Thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά συμφωνεί με τους προλαλήσαντες ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα είναι σίγουρα όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Και μετά την τελευταία δημόσια ακρόαση γίναμε μάρτυρες ακόμη και μιας επιδίνωσης ε, σε πολλούς τομείς πολιτιακών ε, και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και φυσικά εμείς επικεντρώμαστε κυρίως σε οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για να καταμετρήσουμε το βαθμό ανάπτυξης της Κίνας. Αλλά είναι ανησυχητικό αυτό που διαπιστώσαμε την τελευταία διετία, ότι υπάρχει μια μετάβαση της πολιτικής ε, και μία εκτροπή όλο και μεγαλύτερη από τους κανόνες του κράτους δικαίου εκ μέρους της ε, κινέζικης ηγεσία. Αυτό μας προβληματίζει τα μάλα, όχι μόνο γιατί θίγει τις ίδιες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα ζωτικά της ε, συμφέροντα. Πολλές συζητήσεις έγιναν και πολλές συστάσεις υποβλήθηκαν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εκμεταλλευτούμε την εργαλειοθήκη μας, τους μηχανισμούς και το προστάσιο που έχουμε στο διάλογο με την Κίνα και στη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Σίγουρα ο διάλογος είναι το ένα στοιχείο και μάλιστα πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια αξιολόγηση αυτού του διαλόγου με την Κίνα που κατέληξε σε μια σειρά συστάσεων για την αναβάθμιση του διαλόγου αυτού και σας διαβεβαιώ ότι και οι συστάσεις που ακούσαμε προηγουμένως αντικατοπτρίζονται σε αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινήσαμε συζητήσεις με τους Κινέζους ομολόγους μας στη Μαδρίτη και τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις συστάσεις. Και σίγουρα θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τους Κινέζους εταίρους μας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να απαξιώσουμε το διάλογο, γιατί σίγουρα μας δίνει την ευκαιρία δύο φορές το χρόνο να έχουμε βρεθεί συζητήσει με αξιωματούχους της ε, Κίνας και σημαντικούς ε, ηθήναντες για να δούμε πού έχουμε κάποιο κοινό έδαφος ε, και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σημειώνουν τον προβληματισμό μας και η εμπειρία μας έχεις δείξει ότι όταν τα πράγματα λέγονται με σαφήνεια, υπάρχει κάποια βελτίωση από πλευράς της Κίνας και για την κατάσταση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τους συνηγόρους τους και ούτω καθεξής. Επίσης συμφωνώ με την ομόφωνη αυτή έκκληση για ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών εστερνιζόμαστε αυτή την ε, πρόταση και έχουμε και άλλες ιδέες. Γιατί τώρα περνάμε από την κατάσταση πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας σε μία φάση όπου εφαρμόζεται πλήρως η νέα συνθήκη της Λισαβόνας που αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κέριο τομέα δραστηριότητας. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε την πολιτική της πυθούς προς την Κίνα ενθάρρυνσης ε, να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, να βοηθήσουμε την ε, κινέζικη διοίκηση να υιοθετήσει πολιτικές που σέβονται όλο και περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και την κοινωνία των πολιτών της Κίνας για να διεκδικεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματά της. Και εκεί προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μας για μια διεθνή συνένεση ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δείξουμε περισσότερη πυγμή και αποφασιστικότητα απέναντι στο κλασικό επιχείρημα της Κίνας ότι ε, είναι το δικό της συμφέρον να μην ε, να, να διασκεδάσει οποιαδήποτε μας ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναλαμβάνω, έχουμε σημαντικό ε, οπλοστάσιο. Το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημόσιες διακηρύξεις, τις ε, εμπιστευτικέ συνεδριάσεις που έχουμε και που αναλύουμε αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει πάντως να εξασφαλίσουν μια συνέχεια και συμπερίληψη του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στην διάσκεψη κορυφής και αυτό αποτελεί τμήμα της στρατηγική μας. Σα ευχαριστούμε. Πολύ έχετε ακούσει για αυτή την αξιολόγηση του, του Διαλόγου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωση Κίνα. Γιατί λοιπόν δεν το ζητάμε και δημοσίως, γιατί υπάρχει ο κανονισμός 1049 του 2002 για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Οπότε, μια και μας λέει ο κύριος Ρόκας ότι πολλές από τις ιδέες που ακούσαμε στη δημόσια μας ακρόαση από τους καλεσμένους και εμπειρογνώμονές μας αντανακλώνται στο έγγραφο της αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά το βάρος απόδειξης το φέρουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποδειχθεί και τέτοιο, νομίζω ότι δικαιούμαστε να λάβουμε αυτά τα έγγραφα. Δικαιούστε, οπότε μπορείτε να τα ζητήσετε. Σας παραπέμπω στον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού 1049, ο κύριος Στάνοκ. Ευχαριστώ. Είμαι υπερήφανος που είχα δώσει ε, επίσημα και σε μια αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην Κίνα πριν από τρία χρόνια. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και ακούω συνέχεια τα ίδια. Με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και θα με κατηγορούσαν και για μεροληπτικό, γιατί είμαι ε, φίλος οργάνωσης για την Ταϊβάν και είναι ένα πραγματικά εμπορικό θαύμα. Αρχίζει και αναδεικνύεται στην δεύτερη οικονομία παγκοσμίω και σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ε, η Ινδία που είναι μια χώρα που γνωρίζω καλά και την ε, λατρεύω και η Ινδία και η Κίνα επανέρχονται στην πρωτοκαθεδρία που είχαν τον 18ο αιώνα. Ήταν από τις ε, σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, τις τρεις πρώτες οικονομίες του κόσμου. Βέβαια δυστυχώς ε, η πολιτική, της, η πολιτική τους πρόοδος δεν είναι αντάξια της οικονομικής τους πρόοδου. Και οι θύνοντες της Κίνας μου λένε ότι και μόνο από τις διαστάσεις που έχει χώρα αποκλείεται το παραδοσιακό μοντέλο της δυτικής πολιτικής πολυμορφίας. Αλλά έχουμε και άλλες τόσο μεγάλες χώρες και παρόλα αυτά ε, εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες και πολυμορφία. Ε, η Ταϊβάν, για παράδειγμα, και εκεί υπάρχει πλειοψηφία των Χάν και είναι υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Γιατί λοιπόν η Κίνα να μην προχωρήσει προς το δρόμο του εκδημοκρατισμού. Η Ταϊβάν συνεχίζει να υφίσταται απειλές ε, για στρατιωτική εισβολή εκ μέρους Κίνας και παρενοχλείται συνεχώς. Και νομίζω ότι αποκλείστηκε και από διεθνείς οργανώσεις. γιατί κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το, το δόγμα της ενιαίας Κίνας. Πρόσφατα είχαμε τα γενέθλια του Δαλάη Λάμα και πολλοί θηβετιανοί μας εξιστόρισαν ε, τα δεινά τους ε, από την κινέζικη κυβέρνηση. Επίσης ε, συνεχίζονται οι διώξεις πολλών Κινέζων και εφαρμόζεται πολλές φορές η οικονομική δολιοφθορά. Επίσης, ε, περιορίζει εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες σε κάποια στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και μάλιστα ακόμη και προϊόντα από αυτά τα στρατόπεδα έχουν πρόσβαση στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Περιορίζει την ελευθερία έκφρασης ε, στο διαδίκτυο, έχει αποκλείσει το Google και μάλιστα χρησιμοποιεί η Κίνα και εμπορική πίεση, γιατί έχει μεγάλη εγωστική δύναμη, για να εξαναγκάσει ε, εταιρείε όπως τη Utelsat ε, που αναμετέδεκε στους Falun Gong να κλείσουν τις δραστηριότητες εκεί. Και μάλιστα η Falun Gong έκανε ένα, μια εκστρατεία για να παραιτηθούν πολύ από το Κομμουνιστικό Κόμμα και με από την εξτρατεία αυτή 5 εκατομμύρια Κινέζοι επέστρεψαν τις κομμουνιστικές του ταυτότητες. Γι' αυτό και οι Κινέζοι θεωρούνται, η Κινέζικη κυβέρνηση θεωρείται ότι απειλείται από τη Falun Η Κίνα επίσης υποστηρίζει υπόπτα καθεστώτα όπως του Ελέμπασίρ στο Σουδάν ή την ε, στρατιωτική χούντα στη Βερμανία και Επίσης υποστηρίζει και το βάναυσο δημοκρα... Ε, καθεστώς, δικτατορικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας που είναι από τα πιο απολυτερχικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο η Κίνα θα έχει επιρροή για να βελτιώνονταν η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν το κάνει. Η Κίνα με την σημαντική της συνεισφορά στον πολιτισμό διεθνώς και μια χώρα που έχει τόσο ε, πανάρχιο πολιτισμό, ελπίζω κάποια στιγμή να επιτρέψει την ελευθερία και στο λαό τη. Ευχαριστώ και Τάνο και κυρία Λοχμπίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλες τις ομιλήτρες και τους ομιλητές. Ακούσαμε πολλές συστάσεις και πολλές πληροφορίες. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να τις αφημιώσουμε. Χαίρομαι πολύ που ο Λόρδος Τέβερσον του Ηνωμένου Βασιλείου μας είπε ότι στα πορίσματα των εργασιών τους, δεν θεωρεί ότι η οικονομική συνεργασία ε, θα φυγεί εάν κανείς μιλεί ξεκάθαρα για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων με την Κίνα. Στο ίδιο έχουμε στο πλαίσιο των γερμανικών σχέσεων με την ε, Κίνα υπάρχει μεγάλη απήχηση στον τύπο όταν βγαίνει κάποιος κυβερνητικό αξιωματούχο και ε, μιλεί αυστηρά για θέματα ανθρώπινων ε, δικαιωμάτων στην Κίνα. Δεν έχει όμως αυτό, δεν επηρεάζει όμως αυτό τις εμπορικές σχέσεις. Είπατε επίση ότι δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό στην αντιπροσωπεία της Ένωσης που να ασχολείται με θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα. Τώρα με την νέα υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και λόγω ε, του τεράστιου εύρου των σχετικών προβλημάτων στην Κίνα θα είναι ε, σκόπιμο να ενισχυθεί το προσωπικό αυτό. Ο κύριο Γιάν Χάι μα ζήτησε να αναπτύξουμε μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεργασία και αντιμετώπιση της ε, Κοινωνία των πολιτών στην Κίνα. Δεν θα ε, μπω σε όλες τις λεπτομέρειες βέβαια. Σχετικά τώρα με την κριτική που ασκήθηκε ε, στο σεμινάριο της, ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, είναι η δεύτερη φορά που ακούμε σοβαρή κριτική από διάφορες μη κρατικές οργανώσεις, αλλά και συστάσεις για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού αυτού με ξεκάθαρα benchmark, με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για παράδειγμα για την Κίνα να πει η Κίνα πότε πρόκειται επιτέλους να κυρώσει την Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Πολιτικών Δικαιωμάτων που έχει ήδη υπογράψει. Εγώ δεν θέλω να ξανακούσουμε τέτοια κριτική, θέλω να δράσουμε και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κάποιες προτάσεις σχετικά με το πώς θα αντιδράσει στις κριτικές αυτές. Μπόρεσα επίσης να διαβάσω το απόρριτο έγγραφο και νομίζω ότι όντως υπάρχει χώρος για βελτίωση γιατί η αντιμετώπιση των ευρωβουλευτών εγώ ήμουν παλαιότερα μέλος μη κρατικής οργάνωσης και είμαι τώρα ευρωβουλευτής και νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω μάλλον τη λογική ότι κινδυνεύει ασφάλεια εάν έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα. Έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα απορρίτα έγγραφα, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε αρκετή, για ε, αρκετό χρόνο και επίσης να μπορέσουμε να κατήσουμε σημειώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρατε. Θα τονίσω στην, βελτί... στην, συγγνώμη, στην ε, σύσταση που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, βλέπουν μια επιδείνωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συμφωνώ με όσους είπαν ότι ο διάλογος είναι αδιαφανής. Νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε στα όσα προβλέπει τη συνθήκη της Λισαβόνας και να ε, απαιτήσουμε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο διάλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ αναμένω να δω και πιέζω να βγάλει ένα πανό εδώ το Κοινοβούλιο για τον ε, Ουτζά και όλους τους άλλους ε, θαραλέους υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως έχουμε για την Aung San Suu Kyi. Είναι σημαντικό. Επίσης να σημειωθεί, να σημειωθούν μάλλον οι συστάσεις που έκαναν διάφοροι ομιλητές, ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στην ανάπτυξη των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών στην Κίνα. Είτε πρόκειται για ενίσχυση των εκστρατιών που διεξάγουν οι οργανώσεις αυτές είτε πρόκειται για την υποστήριξη των θυμάτων. Θυμούμε που διάβαζα και σε κινέζικα έντυπα, σε κινέζικες εφημερίδες και αυτές που δημοσιεύονται στα αγγλικά με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων το δράμα των γονιών των παιδιών εκείνων που σκοτώθηκαν όταν κατέρευσαν τα σχολεία στον σεισμό του Σετσουάν και που οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν μια απίστευτη καταπίεση γιατί το μόνο που ζητούσαν ήταν να τους αποδοθούν οι σωροί των παιδιών τους. Υποστηρίζω, για παράδειγμα, και τις ομάδες δικηγόρων οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ των δικαιωμάτων των θυμάτων του AIDS, υπέρ ε, των θυμάτων των ε, αναγκαστικών απαλωτριώσεων και σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για τη Tiananmen. Εμείς πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα αυτά και να τα βάλουμε και στον προϋπολογισμό μας σε κάθε οικονομικό μηχανισμό που διαθέτουμε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ε, είναι πολύ σημαντικά όσα μας είπε η κυρία Χόλτσμαν, να υποστηρίξουμε δηλαδή τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και ελπίζω η ΕΦΤΕΛΣΑΤ να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της, διότι υποχώρησε απέναντι στις κινέζικες πιέσεις. Το ίδιο σημαντικό είναι να βγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα από αυτό το γκέτο του διαλόγου των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπουν παντού και να τίθεται και σε κάθε διαπραγμάτευση εμπορικού χαρακτήρα. Εγώ για το λόγο αυτό προτείνω να ζητήσουμε από τον πρόεδρο των εξωτερικών υποθέσεων να κάνει μια κοινή συνεδρίαση με την, με την Επιτροπή Εμπορίου. Τα ανθρώπινα αυτά δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που τόσο υπερηφανεύεται η Κίνα ότι τα έχει προωθήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και είναι αλήθεια αυτό σε πολλές, ε, από πολλές πτυχές, από πολλές απόψεις, αλλά πρέπει να μπουν στον διάλογο τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλες πτυχές, για παράδειγμα και η προστασία των καταναλωτών. Είδαμε το πρόβλημα αυτό με το μολυσμένο γάλα, με τις μολυσμένες οδοντόκρεμες που είναι πολύ σημαντικά για τους Κινέζους, είναι όμως σημαντικά και για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Και... και η Κομισιόν είπε ότι βλέπουμε αυτή τη μετακίνηση πολιτικής που ξεφεύγει από, κράτος δικαίου, από το κράτος δικαίου και τις αρχές του. Πάει και γίνεται η, ε, η Κίνα όλο και περισσότερο η Άγρια Ανατολή ε, χωρίς κανένα νόμο. Πράγματι υπάρχει μεγάλη πρόοδο στην Κίνα την οποία αναγνωρίζουμε σε πολλούς τομείς. Αλλά ε, τι νόημα έχει αυτό χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου. Και το ίδιο για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Αφρική. Όπου γνωρίζουμε ότι υποστηρίζει τον Μπασίρ, την Βυρμανία, το Κονγκό, το καθεστώ στο Κονγκό και το καθεξής. čas, se Εν τέλει, το εξή. Στον τελευταίο διάλογο που κάναμε στη Μαδρίτη το προηγούμενο μήνα, ο Δίος Πάραδα, Αμερικανός εκπρόσωπος, είπε η Κίνα παραπονιέται, η Κίνα καταγγέλει το Γουαντάναμο, αλλά υποφελήθηκε η ίδια. Έστειλε ανακριτές στο Γουαντάναμο. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να θέσουν τα θέματα αυτά. Και τέλος, θα ήθελα να απαντήσει η Κομισιόν στις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Μέτεν για τον διάλογο για στρατιωτικά θέματα. Έγινε ο διάλογος αυτός. Εάν έγινε ο διάλογος αυτός θέλουμε ενημέρωση και να οργανώσουμε κάποια κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο οι Αμερικανοί. Έπαιξε ρόλο ώστε να μην αρθεί το εμπάργο εξοπλισμών. Στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας όταν είχε αναλάβει την δέσμευση η Γαλλική Προεδρία στην αρχή της Προεδρίας της να άρει το εμπάργκο, εν τέλει υποχώρησε λόγω και της αντίδρασης του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Γκόμες. Η Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ και πάλι. Ευχαριστώ που μου δίνεις και πάλι το λόγο. Σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Αφορά